Oui. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει γεμίσει η αίθουσα, λέει ο Πρόεδρος, και μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καταρχήν, να υιοθετήσουμε την ημερησία διάταξη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση. Περνάμε στην έγκριση των πρακτικών Της 23 τετάρτη και 23 Σεπτεμβρίου και της 30 Σεπτεμβρίου 2013. Υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι. Επομένως εγκρίνονται και τα πρακτικά. Για τις ανακοινώσεις τώρα του Πρόεδρου. Θα ήθελα να αναφερθώ στον πέμπτο τριμερή διάλογο για τη ΜΥΦΙΤ που έλαβε χώρα στι 9 Οκτωβρίου. Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα, η διάθρωση των αγορών, διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, προστασία των επενδυτών, πρωτοσύλλες. Και επίση εξετάστηκε και το πεδίο εφαρμογή και οι παρεκκλήσει ε, και ο έκτο τριμερή διάλογο προβλέπεται στι 16 Οκτωβρίου σε ό,τι αφορά την εξυγίανση των τραπεζών. Ο πέμπτο τριμερή διάλογος έγινε στις 8 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Ε, στη συνεδρίαση ολοκληρώθηκαν τα θέματα για το social management και τις συνθήκες τη εξυγίανση και το κείμενο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για το θέμα του Μπεϊλίν τη εξυγίνησης με μέσα συζητήθηκαν βάσει μιας παρουσίαση που έγινε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν δόθηκε εντολή για τις πρόσθετες τεχνικές εργασίες και ο επόμενος τρίμερης διάλογος θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο στις 22 Οκτωβρίου 2013. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Περνάμε επομένως στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το οποίο είναι η έκθεση που αφορά την ασφάλιση έναντι φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Ο κύριος ε, Τέρχο είναι ο εισηγητής και του δίνω το λόγο. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα τις ε, κυρίες αρχές της έκθεσης που βασίζεται στην πράσινη βίβλο που δημοσιεύτηκε την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Και εδώ αναρωτιόμαστε για την αναγκαιότητα ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα αυτό. Κατόπιν θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας παρατηρήσεις και θα περιμένω τις τροπολογίες σας για να είναι συνεκτικό το έγγραφο. Τώρα, όπως γνωρίζετε, τα κράτη-μέλη είναι εκτεθειμένα σε διάφορους κινδύνους και ε, η προβλεψιμότητα των φυσικών καταστροφών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι μετεωρολογικοί και γεωγραφικοί παράγοντες. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάποια προϊόντα που θα ταιριάζουν στην κάθε περίπτωση είναι η καλύτερη λύση για να αντιμετωπίσουν και αυτούς τους παράγοντες. Έτσι λοιπόν υποστηρίζω το να έχουμε ευελιξία ως κύριο στοιχείο για να εγγυηθούμε κάποια προϊόντα ε, που θα ε, ταιριάζουν στην κάθε περίπτωση παρά μια λύση που θα ταιριάζει σε όλους. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της πρόληψης ως το πρώτο βήμα της καταπολέμησης των καταστροφών. Όσο περισσότερο επενδύει κανείς στην πρόληψη, τόσο λιγότερο θα πληρώσει στην περίπτωση που έχουμε κάποια καταστροφή. Επίσης δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την αρχή της ε, ε ατομικής ευθύνης. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι και οι τοπικές κοινότητες να συνειδητοποιήσουν τους υφιστάμενους κινδύνους ε, και το κόστος της έλλειψης προετοιμασίας ε, για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Επιπρόσθετα, η έκθεση τονίζει το ρόλο της ενημέρωσης για να βοηθηθούν οι πολίτες στις επιλογές που κάνουν. Θα είναι χρήσιμο να απτυχθεί ένα δίκτυο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις τοπικές αρχές. Και τέλος, Υπενθυμίζω ότι αφενός οι φυσικές καταστροφές εξαρτώνται από πεντερολογικές ε, και γεωγραφικές συνθήκες και από την άλλη οι ανθρωπογενείς καταστροφές οφείλονται σε λανθασμένη συμπεριφορά ή σε κακή αξιολόγηση των κινδύνων. Έτσι λοιπόν οι φυσικές καταστροφές και οι ανθρωπογενείς καταστροφές καλύπτονται από διάφορα είδη ασφάλισης και δεν θα ήταν σκόπιμο να τα αντιμετωπίσουμε ως ενιαίο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Merci, La parole... Ευχαριστώ κύριε Τέρχο. Για το ΕΛΚ, ο κύριος Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί ε, στην εκθεσή του ανέφερε τα πιο σημαντικά στοιχεία. Πρόκειται για μια πράσινη βίβλο. Η πράσινη βίβλος είναι η πρώτη φάση της εξέτασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν δηλαδή συμφωνούμε με την Κομισιόν ή αν συμφωνεί με την Κομισιόν ότι πρέπει να εξεταθεί το θέμα, ακολουθεί η λευκή βίβλος. Γι' αυτό λοιπόν η πράσινη βίβλος κατά κανόνα είναι ευσύνοπτη. Η έκθεση αναγνωρίζει ότι η αγορά των ασφαλιών είναι ιδιαίτερα ετερογενής, ε, τα κράτη-μέλη είναι εκτεθειμένα σε πάρα πολλούς κινδύνους και υπενθυμίζω την τελευταία έκθεση που έχει υποβληθεί. Υπάρχει η Swiss Ray, η μεγαλύτερη αντασφαλιστική εταιρεία του κόσμου, η δεύτερη μεγαλύτερη και πριν από λίγες ημέρες ανέφερε τους κινδύνους που υπάρχουν από τροπικούς κυκλώνες, από ε, πλημμύρες, από υπερχιλήσεις ποταμών, από σεισμούς και από τσουνάμι. Το συνολικό λοιπόν αποτέλεσμα είναι το εξής. Οι 10 περιοχές του κόσμου που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο ευτυχώς δεν βρίσκονται στην Ευρώπη αλλά εκτός από τη Τόκο Γιοκαχάμα 57 εκατομμύρια, Μανίλα 34,6 εκατομμύρια, Pearl Δέλτα. στην Κίνα 34,5 εκατομμύρια, Ζάκα Κόμπε 32 εκατομμύρια, Τζακάρτα 28 εκατομμύρια. Ναγκόγια στην Ιαπωνία επίσης 23 εκατομμύρια, Καλκούτα 18 εκατομμύρια, Σανγκάι 17, Λος 16 και Τιχεράνη 5,6 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι σημαντικό θέμα αλλά δεν αγγίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε αυτό τον κατάλογο αναφέρονται οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο και αυτή είναι μια ανεξάρτητη μελέτη της Σουίσρε που αξίζει να της ρίξει κανείς μια ματιά. Γι' αυτό λοιπόν στην Ευρώπη όπως αναφέρει και η Πράσινη Βίβλος οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι τεράστιες κυρίως όσον αφορά τους ε, κινδύνους ε, σεισμού ε, και για τις ε, πλημμύρες ε, και εκεί υπάρχουν διαφορές, πόσο μάλλον για υπερχιλής ποταμών. Τσουνάμι υπήρξαν κάποια τέτοια φαινόμενα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν έφτασαν στις διαστάσεις του τσουνάμι που έπληξε τις περιοχές του Ειρηνικού. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα με πολύ μεγάλες διαφορές και ο εισηγητής πολύ σωστά το είπε, δεν μπορούμε να βρούμε μια γενικευμένη λύση για όλες αυτές αυτές τις ε, περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει βοήθεια από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Και στην πρώτη συζήτηση είπα ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ανάληψη ευθυνών. Δεν μπορεί το κράτος να παρεμβαίνει. Το θέμα δεν είναι καλό ή κακό το κράτος, αλλά πρόκειται για φυσικές καταστροφές που κατά κανόνα δεν είναι προβλέψιμες. Εγώ ε, πριν από μερικές εβδομάδες επισκέφτηκα το Τόκιο και επισκέφτηκα και το επίκεντρο του του σεισμού. Στην Ιαπωνία λοιπόν έχουν αναπτύξει ένα σύστημα όπου οι 170.000 ε, σεισμογενείς ε, εκδηλώσεις ε, που υπάρχουν στην Ιαπωνία καταγράφονται μέσα σε δύο λεπτά. Η δημόσια τηλεόραση ενημερώνει για την περιοχή, τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις, αλλά ξέρετε στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παρεμφερές σύστημα. Το σχέδιο της έκθεσης καλεί την Κομισιόν να διασφαλίζει την πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και υπογραμμίζει την ιδία ανάληψη ευθυνών. Ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσεις της αγοράς που να καθιστούν την παρέμβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Λίγο κρίσμα ή κάπως αρνητικά θέματα είναι τέσσερα. Το πρώτον, αναφέρεται ότι ο βαθμός διείσδησης είναι τελείως διαφορετικός στα κράτη-μέλη και αυτό οφείλεται σε πολιτιστικές, γεωγραφικές και άλλες διαφορές. Αυτό όμως πρέπει να συμπληρωθεί. Κατόπιν, ε, στο σημείο υπαριθμών 8. Εκεί καλείται η αγορά των ασφαλιών να προσφέρει προσιτή ε, προστασία και κίνητρα για τους ε, πολίτες και εκεί πρέπει να διευκρινίζεται ποια μπορεί να είναι αυτά τα οικονομικά κίνητρα. Σημείο υπαριθμών 9. Καλεί τις ασφαλιστικές εταιρείες ε, να διαμορφώσουν απλούστερες ε, τις συμβάσεις. Ε, θα ήθελα στην κυρία Περές να απευθυνθώ εδώ, η οποία θέλει να συμπεριλάβει και τις παροχές ασφαλιών από τον τομέα BRIPS. Νομίζω ότι αυτές τις πληροφορίες πρέπει να τις ρυθμίσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να περιλαμβάνονται σε απλά εγχειρίδια. Γιατί το να προβλέψει κανείς ένα σεισμό ή ε, ένα τσουνάμι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Σημείο υπαρθμών 13. Ναι μεν αναφέρει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ιδία ανάληψη ευθυνών εκ μέρους των πολιτών. Εδώ όμως τίθεται το ερώτημα τι ακριβώς εννοούμε. Και ίσως θα πρέπει να διευκρινίσουμε στον εισηγητή τι ακριβώς επιθυμούμε στην άδελφη. Ίσως αυτός να έχει κάποιους ε, περισμούς ε, λόγω της μορφής της έκθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την έκθεση αυτή τη βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμη για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τόρβαλτς. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του όπως είπε ο κύριος Λάγκεν, και εγώ συμφωνώ με τα περισσότερα από τα σημεία της έκθεσης. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της πρόληψης και της ενημέρωσης, συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα. Μία μεγάλη πρόκληση για τις ασφαλιστικές και τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι ότι δεν έχουν αρκετά δεδομένα για τους κινδύνους που έχουν οι φυσικές καταστροφές και αυτό σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολο για αυτές να παρουσιάσουν την καλύτερη μορφή ασφάλισης στην κατάλληλη τιμή για την ε, σωστή καταστροφή. Είπε ο εισηγητής ότι δεν είναι καλή μία ταιριάζει σε όλους και συμφωνώ. Από όσο ξέρω, πολλά κράτη-μέλη έχουν διάφορα συστήματα που λειτουργούν σήμερα και δεν ε, φαντάζομαι γιατί να θέλαμε να απομακρυνθούμε από αυτές τις λύσεις. Και επίσης η αντασφάλιση είναι ε, παγκόσμια και ε, έτσι ε, έχουμε κάποια ασφάλιστρα τα οποία μπορεί να, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν αντιρρήσεις για το υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης ακόμη και αν φαίνεται απαραίτητο να μειώσουμε το κόστος των ασφαλίσεων, πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα κίνητρα πίσω από τον υπάρχει ασφάλιση και ε, το έργο επίσης να αποτρέψουμε τις πιθανές καταστροφές είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης ε, ε, έχουμε στο ίδιο έγγραφο να, αντιμετωπίζονται και οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς καταστροφές σε μια ανθρωπογενή καταστροφή, κάποιο έχει πάντοτε την ευθύνη, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τι φυσικέ καταστροφέ. Έτσι λοιπόν, οι φυσικέ καταστροφέ από μια σκοπιά ασφάλιση πολλέ φορέ αντιμετωπίζονται ε, στο πλαίσιο τη ε, ασφάλεια τη ιδιοκτησία, ενώ ανθρωπογενεί καταστροφέ από την ασφάλεια ευθύνη. Ε, είδαμε και τι έγινε στη Φουκοσίμα, όπου φυσικέ καταστροφέ τροποποιήθηκαν ε, σε ανθρωπογενή τις ε, καταστροφές ε, και ε, είδαμε ότι μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες ζημίες από τα νερά. Και σε ό,τι αφορά την ευθύνη, ξέρω ότι η Κομισιόν εργάζεται για μια οδηγία για την ευθύνη στις φυσικές καταστροφές και υπάρχει και μία οδηγία που αφορά την ευθύνη σε περίπτωση πυρηνικών ε, ατυχημάτων. Έχουμε λοιπόν πολλές γενικές διευθύνσεις στην Κομισιόν που εργάζονται επί του θέματος αυτού και αναρωτιέμαι αν ε, τελικά θα καταλήξουμε σε ένα κανονισμό αντιφατικό και ε, μάλλον αυτό αν καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο θα έχουμε μια γραφειοκρατική καταστροφή που θα την έχει προκαλέσει η Κομισιόν. Ο κύριος ε, Λάγκεν ότι είπε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και μαζί του και με τους υπόλοιπους και τις συζητητές με ένα πολύ συνεκτικό τρόπο. Και σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δω τώρα. Ποιος αντικαθιστά την κυρία Ίτσι, θέλετε να πάρει το λόγο αμέσως. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι όμως συντομότατος. Εκπροσωπώ την συνάδελφό μου Μιτσίτη ότι δεν μπορεί να προσέλθει σήμερα. Κολλείεται. Αναφέρεται βέβαια όπως ξέρετε στις ε, ανθρωπογενείς και μη καταστροφές. Το κείμενο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και συμφωνεί, λέει η συγκήτρια, η συνάδελφός μου, με τον εισηγητή ότι δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη προσέγγιση για όλες τις περιπτώσεις, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν τελείως άχρηστο. Η πρόληψη και η πληροφόρηση είναι το καλύτερο. Υπάρχει συμφωνία γενικά ότι η πρόσβαση σε περισσότερη πληροφόρηση This information, however, should Για να πληροφορείται καλύτερα ο καταναλωτής έτσι ώστε να έχει αυτός την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Η έκθεση όμως, η έκθεση όμως λέω, έχει και μερικές ελλείψεις. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε και την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ κυβερνήσεων και καταναλωτών χωρίς να ξεχνάμε και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για την πρόληψη νομίζω ότι η έκθεση πρέπει να τονίσει περισσότερο τη σημασία που έχουν οι κρατικές αρχές για την πληροφόρηση των πολιτών. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η έκθεση το λέει, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα, πολλά περισσότερα. Και ιδιαίτερα να αναφέρεται το γεγονός ότι are occasions when on those indeed make ότι δηλαδή πρέπει να αποφύγουμε τη χειροτέρευση των καταστάσεων. Και να γίνονται όλα αυτά απλούστερα. Αυτό συνδέεται και με το θέμα της πληροφόρησης. Η ασφαλίσεις πρέπει να βασίζονται στην αποτίμηση του κινδύνου. Για να είναι αποτελεσματικές χρειάζεται δε επαρκής πληροφόρηση. πληροφόρηση. Πιστεύω ότι το θέμα του ηθικού κινδύνου δεν έχει εξεταστεί επαρκώς. και επίσης νομίζω ότι Insurance. ότι αυτό πρέπει να ισχύει και για τις υποχρεωτικές και για τις μη υποχρεωτικές ασφαλίσεις. Για τις υποχρεωτικές συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι η ασφάλιση για τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές δεν είναι τελείως απαραίτητη. Γι' αυτό προτείνουμε, θα, θα υποβάλουμε τροπολογίες σχετικό σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ο κύριος Ζαμπολής. Ευχαριστώ κύριε Ζαν Πολ Γκοζές μου. Θα ήθελα να πω προς τον κύριο Σαμποτέρο ότι η έκθεσή του έχει δύο πλευρές. Μία που τη βρίσκουμε πολύ θετική είναι η πρόληψη και η πληροφόρηση και μία που μας φαίνεται πιο συζητήσιμη και που είναι το θέμα της ατομικής ευθύνης έναντι της κρατικής διάφτης. Οι συνάδελφοι θεωρούν ότι χρειάζεται καλύτερος ορισμός των θεομηνιών από τις ανθρωπογενείς. Αλλά αυτό είναι δύσκολο και ακριβώς η ευθύνη του ανθρώπου είναι όλο και σημαντικότερη και για τις θεομηνίες, δεν μιλάω για τους σεισμούς βέβαια και τα παλιραϊκά κύματα, αλλά για τις πλημμύρες, για τα κύματα θερμοπληξιών λοιπά. Γίνεται λοιπόν εδώ ένας αγώνας δρόμου καταστροφισμού. Τώρα για την ίδια την έκθεση το ότι τονίζει περισσότερο την ε, πρόληψη μας φαίνεται κάτι θετικό διότι οι καταστροφές πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται και το κόστος της αντιμετώπισης τους γίνεται όλο και βαρύτερο και μπορεί να υπονομεύσει ολόκληρη την ανάπτυξη κάποιας περιοχής ή χώρας ή και του συνόλου του πλανήτου. Άρα όλα αυτά για την πληροφόρηση και την παιδεία για αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά. Αλλά πρέπει να απλοποιηθεί, να απλοποιηθούν τα πράγματα για τα άτομα που αντιμετωπίζουν ξαφνικά μια τέτοια καταστροφή. Να τους βοηθήσουμε δηλαδή σε επανενωσιακό επίπεδο γράφοντας νομοθετήματα τυποποιημένα απλά και άμεσα για να γνωρίζουν και αυτοί τι κίνδυνος καλύπτεται από την νομοθεσία και τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε και τη δημιουργία ενός μιας ιστοσελίδας, ενός ιστοτόπου με τις πληροφορίες αυτές, όπου να μπορεί ο καθένας με ένα κλικ να πάνω στην περιοχή ή την πόλη του ή το χωριό του ή τη γειτονιά του ή το σπίτι του ή το παράθυρό του να βλέπει τι κίνδυνοι υπάρχουν. Να ταυτιστούν λοιπόν οι κίνδυνοι ώστε δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση μας φαίνονται σωστά πράγματα αλλά και όμως οι διαφορές που έχουμε με τον εισηγητή αφορούν κυρίως το ύφος γιατί νομίζουμε ότι τονίζει ιδιαίτερα την ατομική ευθύνη και τη διαχωρίζει από το ρόλο του κράτους και κάποιας πανενουσιακής πιθανής παρέμβασης ενώ η καταστροφές και θεομηνίες αυτές ξεπερνούν κατά πολύ το ατομικό πλαίσιο και το εθνικό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένα προϊόντα ασφαλιστικά για την κάθε κατηγορία θεομηνίας, αλλά πρέπει η Ευρώπη να καθορίσει στόχους ένα γενικότερο πλαίσιο σύγκλησης που να επιτρέπει ακριβώς να ασκείται ευκολότερα η ατομική ευθύνη, να γίνει κάποια εναρμόνιση όχι μόνο για την παιδεία αλλά και για όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια για να γνωρίζουμε τι ακριβώς αναλαμβάνει το κάθε άτομο όταν υπογράψει μια τέτοια ασφάλιση. Για τις ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως οι χημικές μολύνσεις, τα πυρηνικά ατυχήματα, εδώ τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ αυστηρότερα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ισχύει, δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας ποτέ πλήρως να ασφαλίσει ατυχήματα σαν τα πυρηνικά. Και γι' αυτό θα καταθέσουμε τροπολογίες. Και θα συνεργαστούμε βέβαια με όλους τους σκιώδεις και με τον ίδιο τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίνπο αντικαθιστά τον κύριο Φόξ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Φόξ μου ζήτησε να πω ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με την έκθεση για τις φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα χαίρεται ιδιαίτερα που αναφέρει ο συγητής ότι οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο τσουβάλι γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικά φαινόμενα με διαφορετικές ε, ευθύνε και διαφορετική αστική ευθύνη. Ο κύριος Φόξ επίσης πιστεύει ότι στον τομέα αυτό δεν υπάρχει στρέβλο της αγοράς που να αιτιολογεί την παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χαίρεται που ο εισηγητής δεν πιστεύει ότι μια γενικευμένη προσέγγιση ταιριάζει σε αυτό τον τομέα. Συμφωνεί με τον εισηγητή ότι ένα μη υποχρεωτικό πλαίσιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξουμε προϊόντα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Βέβαια ο κύριος Φόξ ανησυχεί λιγάκι σχετικά με την τυποποίηση γιατί αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα και διαφορετικοί ορισμοί και είναι αδύνατο να υπάρξουν γενικευμένα στάν Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Φόξ καλεί τους συναντέλφους του ε, να παρουσιάσουν και να επιμείνουν σε μια ρεαλιστική προσέγγιση, κάτι που υπήρξε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι όπως είπαν και οι άλλοι ομιλητές η έκθεση του συναδέλφου ε, αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε σοβαρά διότι ε, ε, θέτει σοβαρά ζητήματα. Το λέω αυτό γιατί έρχομαι κάτω από το κράτος μιας χτεσινής σεισμικής δόνησης που έγινε δυτικά της Κρήτης, νομίζω ότι η γεωγραφία τη γνωρίζετε, είναι, ναι, είναι η περιοχή που έχει δώσει το μεγαλύτερο σεισμό πριν από χρόνια βέβαια, στη Μεσόγειο, που είχε δώσει και το μεγαλύτερο τσουνάμι, όπως λένε τα πράγματα. Και εξ αυτού υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία γιατί το ανέφερα αυτό. Σωστά πρέπει να ξεχωρίσουμε τα αίτια σε φυσικά αίτια και ανθρωπογενή. Αλλά τα φυσικά αίτια δεν είναι όλα το ίδιο πράγμα. Άλλο πράγμα, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, είναι ο σεισμός. Δυστυχώς ούτε στην Ιαπωνία ούτε στη χώρα μου που είναι σεισμογενείς χώρες έχει βρεθεί τρόπος να τον προβλέπει στο σεισμό. Και άλλο πράγμα είναι οι πλημμύρες, οι κατακλυσμοί και άλλα φαινόμενα τέτοια που έχουν προκληθεί όπως αναγνωρίζει και η πράσινη βίβλος της Επιτροπής από τις κλιματικές αλλαγές επομένως από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο περιβάλλον. Και αν είναι κάτι να ερευνηθεί αν και είναι γνωστό αυτές οι πολιτικές που βλάπτουν το περιβάλλον και στη συνέχεια επηρεάζουν πια το κλίμα πρέπει να αλλάξουν. Επομένως ως προς αυτή την κατηγορία των φαινομένων Νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά και δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε και εννοώ την Επιτροπή η οποία δεν τα, δεν τα συγκεκριμενοποιεί αυτά τα ζητήματα. Δεύτερο, υπάρχουν ε, βεβαίως και οι ανθρωπογενείς ε, παρεμβάσεις που δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα, προφανώς η πρόληψη, εδώ συμφωνώ με τον εισηγητή και ο καθένας θα ε, συμφωνήσει, ε, και η ενημέρωση είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Αναφέρομαι ε, ίσως φλιαρώντας ε, παραπάνω, ας πούμε πρόληψη από τους σεισμούς, τι, ποια μπορεί να είναι. Τα κτίρια να χτίζονται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, ούτως ώστε οι επιπτώσεις από ένα σεισμό που δεν μπορείς να το σταματήσεις, να είναι ε, οι λιγότερες δυνατές, να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Για άλλες μορφές φυσικών φαινομένων, η ενημέρωση πώς αντιδράς, προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως εδώ αν μπορεί να καθιερωθούν θεσμοί ανταλλαγής εμπειριών για να ενισχύσει το σκέλος της πρόληψης είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Μια τρίτη παρατήρηση, γενικές θα είναι οι παρατηρήσεις και θα τα συγκεκριμενοποιήσουμε τις προτάσεις μας με τροπολογίες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν σαν στόχο την προστασία των πολιτών καταναλωτών από αμφιλεγόμενα και ζημιογόνα πακέτα ασφάλισης. Να το πω διαφορετικά, ε, επειδή σε αυτό το τομέα υπάρχει μια τάση να αυξηθεί επειδή αυξάνονται τα φαινόμενα είτε από τη μια αιτία είτε από την άλλη αν δεν υπάρχουν κανόνες αυστηροί κανόνες όσον αφορά, όσο αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες φοβάμαι κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι ότι μπορεί να φτιαχτεί μια φούσκα, πιθανή φούσκα στην αγορά ασφαλίστρων όπως το είδαμε στο παρελθόν για άλλα βέβαια θέματα. Επομένως αυτό το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου πρέπει να εντοπιστεί. Τέλος, όσο αφορά τις ανθρωπογενείς καταστροφές, νομίζω οι κανόνες ασφαλείας και οι πολιτικές που τις ξέρουμε ότι έχουν επιδράσεις δυσμενείς ε, και στο περιβάλλον και στους ανθρώπους νομίζω ότι πρέπει και να αποφεύγονται και να αποτρέπονται ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και μπαίνουμε στην υπόθεση πώς θα γίνει η ασφάλιση και πώς θα ε, αποφύγουμε φούσκες στα ασφάλιστρα πράγμα που σημείωσα εδώ. Αυτές είναι ορισμένες γενικές παρατηρήσεις. Σε επιμέρους θέματα θα καταθέσουμε τροπολογία. Ευχαριστώ τον εισηγητή που άνοιξε το θέμα και μας έβαλε να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε και να κάνουμε προτάσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Χουντή. Κύριε Λάγκεν, θέλετε να επανέλθετε. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Θα ήθελα να μου επιτρέπετε να συμπλώσω κάτι μετά από αυτά που είπε ο κύριος Χουντής. Κοιτάξτε, η πρόληψη στα κτίρια και για την περίπτωση των σεισμών, κατά την άποψή μου αυτό είναι καθαρά εθνικό καθήκον. Δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι Υπάρχουν ε, κάποιες ε, συμφωνίες ε, που έχουν υπογραφεί, αλλά επειδή δεν υπάρχουν ενιαίες λύσεις, τελικά θα καταλήξουμε απλά σε διόγκωση της γραφειοκρατίας. Η διεθνή συνεργασία, η παρέμβαση, η πρόληψη, σε ορισμένες περιπτώσεις όλα αυτά είναι πολύ λογικά, αλλά δεν είναι δυνατόν επειδή υπάρχει αυτή η χήμερα του κλιματικής αλλαγής ε, να θέλουμε να καταλήξουμε σε γιγαντιαία προγράμματα. Αυτό δεν μπορεί να είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πέμπτη έκδοση της ε, Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τις κλιματικές αλλαγές είπε ότι στην ακραία περίπτωση μέχρι το 2000, ε, μέχρι το 3.000 περίπου ε, θα έχει ανέβει η στάθμη της θάλασσας περίπου το πολύ κατά 15 εκατοστά ε, μάλλον λιγότερο και στην Ευρώπη εξ όσων γνωρίζω αυτό δεν θίγει καμία χώρα άρα δηλαδή δεν πρέπει τώρα να δημιουργήσουμε νέα προγράμματα ενίσχυσης και να χορηγούμε επιδοτήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη αλλά με άλλες χώρες του κόσμου η Κομισιόν θέλει το λόγο, αν όχι, να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ. Δεν θέλει η Κομισιόν. Έχετε το λόγο κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους κοιόδες για τη συνεισφορά τους βλέπω ότι έχουμε μια κοινή προσέγγιση επί του θέματος, επομένως θα είναι καλή και συνεργασία μας όταν ε, στο μέλλον θα διατυπώσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε να εκπονήσουμε το τελικό έγγραφο. Επομένως είμαι αρκετά αισιόδοξο για το αποτέλεσμα αυτού του εγγράφου και πάλι σας ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα. μια κατάθεση τροπολογιών 22 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η συζήτηση για τις τροπολογίες 25 και 26 Νοεμβρίου στη συνεδρία της Επιτροπής και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 17 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια προβλέπεται για το Φεβρουάριο του 2014. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο της της διάταξης, ε, το εξαντλήσαμε, ίσως εσείς να μην εξαντληθήκατε αλλά θα διακόψουμε μέχρι τις 4 για να περάσουμε στο θέμα που αφορά τον ενίο μηχανισμό εξυγίανσης και την έκθεση της κυρίας Φερέιρα. Διακόπτουμε μέχρι τις 4.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 Um, Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Βλέπω ότι όλοι οι κύριοι πρωταγωνιστές είναι εδώ. Επομένως θα προχωρήσουμε και θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης της Ελίσσα για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Θα δώσω λοιπόν απευθείας το λόγο στην Ελίσσα. Ευχαριστώ Σάρων. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να πω πως αυτή η νομοθετική πρόταση για την ε, εξυγίανση των τραπεζών έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο μέτρο που εργαζόμαστε ταυτόχρονα και επί του κειμένου αυτού για την εξυγίανση και παράλληλα με αυτό Εργαζόμαστε επί του κειμένου οδηγίας που θα εφαρμοστεί στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ε, εξυγίανση των τραπεζών. Επομένως, ε, μιλάμε για μία ενιαία εξυγίανση και δεν είναι ένα είδος ε, σφαίρας που περιλαμβάνεται σε μία άλλη ευρύτερη σφαίρα. Εμείς μέχρι τώρα δεν είχαμε επιλέξει να υποβάλουμε τροπολογίες για το κείμενο του ενιαίου μηχανισμού και θα το αναφέρω στο SRM. Στον ε, SRM, ε, στο μηχανισμό αυτό, αποφασίσαμε να μην εισαγάγουμε τροπολογίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ε, κάποια σύγκρουση με το νομοθετικό κείμενο, επί του οποίου εργαζόμαστε στον τριμερή διάλογο και θεσπίζει τους κοινού κανόνες για το τρόπο εξυγίανσης ενός τραπεζικού ιδρύματος. Η κύριες γραμμές μας δεν φύγουν θεμελιώδεις πτυχές της πρότασης όπως έχει υποβληθεί. Μας φαίνεται ότι γενικά η πρόταση της Κομισιόν είναι φιλόδοξη και οδεύει προς την κατεύθυνση που είχε ζητήσει ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 και περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία και σε σχέση με τα οποία μας ενδιαφέρει να μην χάσουμε τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί και απλώς ε, θέλουμε να βελτιώσουμε ή να διορθώσουμε κάποια στοιχεία. Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι το θέμα της απόφασης να τεθεί μια τράπεζα σε διαδικασία εξυγίανσης, όπου, όπως είπα και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, και έχουν κατευθυνθεί τροπολογίες και νομίζω ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν προκειμένου να διευκρινιστεί ότι οι οντότητες είναι αυτές που μπορεί να, είναι οι οντότητες που μπορεί να δηλώσουν ότι ένα τραπεζικό ίδρυμα, ένα χρηματοστατικό ίδρυμα είναι σε στάδιο πρώτης χρονοκοπίας και πρέπει να μπει σε στάδιο εξυγίανσης. Νομίζω ότι αυτή η διευκρίνηση είναι σημαντικό στοιχείο για να έχουμε ε, μία ε, ασφάλεια δικαίου στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και όσοι είναι αντικείμενο της εποπτείας ε, να γνωρίζουν ποια είναι τα κριτήρια που μπορεί να τους θέσουν σε ένα τέτοιο στάδιο προεξυγίανσης και ποιοι είναι οι μηχανισμοί άμυνας έναντι της διαδικασίας αυτής. Έτσι λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι στο επίπεδο εποπτείας θα πρέπει να επικεντρωθεί αυτή η διαδικασία αν και δεχόμαστε ανταλλαγές ε, απόψεων και ευνοούμε να υπάρχουν ανταλλαγές διάφορων απόψεων στα πλαίσια της οντότητας. Όμως πρέπει να ξέρουμε ποιος λαμβάνει αυτή η πρωτοβουλία της σε Ένα δεύτερο σημείο το οποίο μου φαίνεται σημαντικό να υπογραμμίσω είναι το εξής το θέμα της συμμετοχής αυτού του Κοινοβουλίου, όπως έχουμε πράξει είτε στο διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των ε, αρχών εποπτείας, αυτό που και εδώ υπερασπίζουμε για τον ενίο μηχανισμό εποπτείας είναι και εδώ να υπάρχουν κάποιες αρχές ε, που θα διέπουν την επιλογή του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, να υπάρχει δημόσια διαφάνεια και έλεγχος ε, της ε, διαδικασίας από το Κοινοβούλιο. Ένα τρίτο σημείο, το οποίο είναι θεμελιώδες να συζητήσουμε, είναι ύπαρξη ενός ε, μέσου δανειοδότησης ή ενός ε, είδους δημοσίου backstop για να λειτουργεί αυτό το Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο θα πρέπει να είναι λειτουργικό όταν θα τεθεί σε ισχύ και η νομοθεσία. Είναι ένα θέμα πολύπλοκο και σε σχέση με το οποίο το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δώσει ποια είναι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτού του μηχανισμού, αλλά θέλουμε μια αξιόπιστη διαδικασία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 10 χρόνια συνεισφορών μέχρι να έχει τους απαραίτητους πόρους του Ταμείου για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει ένα, μια οντότητα εξυγίανσης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μέσο το οποίο δεν ε, θα χρησιμοποιεί χρήματα από τους φορολογούμενους, αλλά θα πρέπει να επιστρέφονται τα κονδύλια και θα έχουμε συνεισφορές από την ίδια την τράπεζα, από τους ίδιους τους εποπτευόμενους στο ταμείο αυτό. και αυτές οι συνεισφορές επομένως θα γίνονται βάση του κινδύνου και θα πρέπει τα χρήματα αυτά να προέρχονται από την τράπεζα και όχι από τους φορολογούμενους, να μην βγαίνουν από την τσέπη των φορολογούμενων. Και υπάρχει εδώ και ένα άλλο στοιχείο που έχει πολύ μεγάλη σχέση με τον Μπελίν, με τη διάσωση με ίδια μέσα, τα οποία το συζητάμε στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση. Εδώ θα θέλουμε να έχουμε ένα μηχανισμό πυροδότησης, ενεργοποίησης του Ταμείου, αμέσως όταν οι καταθέσεις αρχίζουν να είναι η επόμενη ε, κατηγορία που θα χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση με ίδια μέσα. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά προϋποθέσεων παρέμβασης του τεμείου, προβλέπεται μια σειρά συνθήκων στην νομοθεσία, μια σειρά προϋποθέσεων και θέλουμε να δημιουργεί ασφάλεια στην αγορά, ένα τέτοιο μηχανισμός πυροδότηση. Και θα πρέπει αυτό να γίνεται τη στιγμή που η διαδικασία του Μπέιλιν, της διάσωση με ίδια μέσα, αρχίζει να φύγει τις καταθέσει. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε λεπτομερώς τα διαφορετικά καταθέσεων στο πλαίσιο αυτό, όμως εδώ θέλουμε να υπάρχει μία σύνδεση ότι η παρέμβαση του Ταμείου με δυνατότητα μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων ε, θα πρέπει να πυροδοτηθεί όταν αρχίζουν να θίγονται οι καταθέσεις. Και ένα τελευταίο σχόλιο, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Αφορά το θέμα της ημερομηνία της θέσεως ισχύει όλης αυτής της νομοθεσίας γιατί ο SRM, η για την ανάκαμψη και την εξυγίανση, το Ταμείο και η δυνατότητα της διάσωσης με ίδια μέσα είναι όλα κομμάτια ε, του ίδιου παζλ και θα πρέπει όλα αυτά να είναι συμβατά μεταξύ τους έτσι ώστε να μην διαταραχθεί και η εσωτερική αγορά με τη θέση σε ισχύ όλες αυτές της νέας νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία εγώ κατά κάποιο τρόπο τα είχα αναφέρει και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αυτή τη στιγμή έχει, έχουν καταθέσει και συνάδελφοι τις τροπολογίες. Εγώ θέλω να ενημερώσω ότι και εγώ θα κάνω κάποιες πρόσθετες τροπολογίες, αλλά που δεν αφαιρούν και δεν φύγουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, τις κύριες θεμελιώδεις γραμμές που ανέφερα και μέσω των τροπολογιών ελπίζουμε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να σας πω. Uh, Ευχαριστούμε πολύ για το ΕΛΚ τώρα. Ευχαριστώ πολύ και την Ελίσσα για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας και εκτιμώ ιδιαίτερα την αφοσίωσή μας και των δύο για να διεκπαιρεωθεί το θέμα γρήγορα. Βέβαια η ποιότητα είναι το πρώτο κριτήριο. Υπάρχει γενικά συνένεση ότι ο μηχανισμός αυτός θα είναι ένα από τα θεμέλια της Τραπεζικής Ένωσης και γι' αυτό το Κοινοβούλιο θέλει να καταλήξουμε συμφωνία πριν τις ευρωεκλογές και συμφωνώ και εγώ με αυτό προσωπικά. Βεβαίω χρειάζεται συνεργασία και επομένως πρέπει να δούμε τι θα πράξει και το Συμβούλιο. Συμφωνώ με την Ελίσσα ότι η κατεύθυνση που πήρε βασικά με την πρόταση της Κομισιόν είναι σωστή. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να πείσουμε και το Συμβούλιο. Δεύτερον, Επίσης σημαντική αρχή είναι όπως έγινε για τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας και στην BERT, όπου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει. Αυτά όλα δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε όλα από την αρχή, αλλά να αρχίσουμε από τα συμπεράσματα. Βέβαια δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις για την Μπέρντα, αλλά αν θέλουμε να πράξουμε έτσι πρέπει έτσι να κάνουμε και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι έχω την εντύπωση ότι είναι και θέμα ισοτιμίας εδώ πέρα Ίσως μια τροπολογία να αντιφάσκει με τη γραμμή αυτή που είπαμε για την Bird Για το ευρώ στο πεδίο εφαρμογή ε, συμφωνώ να καλύπτει όλες τις τράπεζες. Το ίδιο κάναμε και για το SSM. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι θα γίνει με τις μικρότερες τράπεζες που δεν είναι τμήμα του Asset Quality Review. Πριν να εξετάσουμε το SSM και το SRM πρέπει να δούμε τι γίνεται με όλες τις τράπεζες. Αλλά ιδιαίτερα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι μικρότερες. Πού πρέπει και αυτές να συμβάλλουν στο Ταμείο με τον κατάλληλο τρόπο αναλογικά. Δεν το ξέρουμε αυτό προς το παρόν. Έπειτα, ο ρόλος της Κομισιόν συζητήθηκε ήδη, αλλά υπάρχει και του Συμβουλίου. Είπαμε να μειωθούν κάπως οι διακριτικές της ευχέρειες, αλλά Υπάρχει το νομικό υπόβαθρο που είναι δεδομένο. Πρέπει όμως να έχει, να ισχυρότερο ρόλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό είναι σίγουρο, για να είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει διενοσιακός ρόλος. Άρα να μην δούμε μόνο τη σύνθεση του Συμβουλίου. Γιατί εγώ θέλω και η, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Κομισιόν να παίζουν ένα ρόλο και καλό θα ήταν να τον αναλάβουν, να παίζουν ένα ρόλο στο Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως ο στόχος είναι το κοινοτικό και όχι το εθνικό συμφέρον. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα καθήκοντά του, αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε άλλη φορά σε περισσότερες λεπτομέρειες. Για το Resolution Fund, είναι προφανές ότι πρέπει να θέσουμε σαν, πρώτα σαν όρο να καταλήξει το SRM. Δύσκολο πολιτικά το θέμα, αλλά πιστεύω ότι, ότι η Ευρωζώνη, το Eurogroup συμφωνεί Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω. Ο απόρριτος χαρακτήρας. Τα σχέδια που θα υποβάλουν οι τράπεζες θέλει το Συμβούλιο να τα συζητήσει το, το Συμβούλιο στην Ολομέλειά του. Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα ήταν σωστό γιατί υπάρχουν εδώ επιστευτικές πληροφορίες που έτσι θα γνωστοποιηθούν δημόσια. Πρέπει να γίνει καλύτερη κατανομή λοιπόν των καθηκόντων μεταξύ της διοικητικής δουλειάς του Συμβουλίου αυτού και της Ολομελίας του. Ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια γρήγορη πρόοδο αλλά και για μένα και για την Κομισιόν και για τη γραμματεία της Επιτροπής μας πρέπει να δούμε πώς θα το συνδυάσουμε όλο αυτό με το θέμα της Μπέρντ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Σίλβη δεν μπόρεσε να γιατί γι' αυτό μου έδωσε τι σημειώσει της για να τις ε, διαβάσω και μιλώ βέβαια και εξ ονόματός μου, αλλά αυτό θα το κάνω αργότερα, αφού έχουν μιλήσει πρώτα οι εκπρόσωποι των εισηγητές. Εκ μέρους των φιλελευθέρων η Σίλβη λέει ότι καλωσορίζει την πρόταση, βεβαίως χρειαζόταν επιγόντως και είναι πολύ σημαντικό ο μηχανισμός ε, να είναι υπόλογος και εκείνη επιθυμεί να συμφωνήσει με τους ε, μηχανισμούς που προβλήπονται στον SSM και πρέπει να επαναληφθούν στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίωνσης, ε, στον SRM. Επίσης αναφέρεται στο ότι το SSM και η BRD πρέπει να είναι υγιείς μηχανισμοί ε, κατόπιν τούτου ε, πρέπει να καλύπτονται από... Ε, πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ μου. Επίσης, ε, θα πρέπει να είναι σαφείς οι αρμοδιότητες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπάρχει περιθώριο ε, ελιγμών. Ε, αυτό είναι πολύ μεγάλο όσον αφορά την Επιτροπή και οι εκ των προτέρων εισφορές εκ μέρους των θεσμών υπάρχουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για να αρχίσει να ισχύει ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης. Η λύση που θα αναζητηθεί θα πρέπει να βασίζεται στη δικαιοσύνη και όλα τα μετέχοντα κράτη ε, θα πρέπει να συμβάλλουν ε, κατά κάποιον τρόπο. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο ψηφοφορίας, ο επόπτης ε, θα πρέπει να είναι παρατηρητής χωρίς να έχει δικαίωμα ψηφοφορίας. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στους φιλοξενούμενους ε, και στους ε, γηγενείς μηχανισμούς, οι επενδύσεις ε, θα πρέπει να γίνονται σε κεφάλαια με υψηλή αξιοπιστία και τομεακά και να υπάρχει και γεωγραφική διαφοροποίηση. Η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει να είναι περιεκτική, να υπάρχει κάποια λύση ε, ανάμεσα στο τραπεζικά δάνεια και την ε, πτώχευση. Στην παράγραφο 4 προβλέπεται το δικαίωμα της αρνησικυρίας, αλλά αυτό θα πρέπει να πάψει να υπάρχει, γιατί δεν είναι απαραίτητη η υποστήριξη, η δημόσια υποστήριξη. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι ο νέος μηχανισμός εξυγίανσης ε, θα μπορεί να συστήνει συμβουλευτικές επιτροπές, γιατί είναι απαραίτητες αυτές οι ειδικέ γνώσεις. Αυτές είναι κάποιες κάποιες ε, έτσι παρατηρήσεις ε, και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στους ε, πράσινους. Ο Σβέν έχει το λόγο. Ο Φιλίπ που είναι συνεισηγητής μαζί μου εξακολουθεί να ψηφίζει την Ήτρε. Καταρχήν θέλω να πω ευχαριστώ πολύ την Ελίζα για την έκθεσή της. Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα την Επιτροπή που προτείνει αυτό το, αυτή την έκθεση και που προτείνει να προχωρήσουμε γιατί αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο έτσι ώστε ο ε, ενιαίος μηχανισμός, ε, ο μηχανισμός στήριξης, ε, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί. Είναι σαφές ε, ότι βρισκόμαστε σε κάποια στιγμή έχουμε φτάσει στο να πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Γιατί ο εποπτικός μηχανισμός, αν δεν υπάρχει ένα κοινό σύστημα εξυγίανσης, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. Και κατ' ουσίαν αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι είναι αυτό το κοινό backstop. Εδώ η Κομισιόν δίνει κάποια απάντηση ακόμα και για προβλήματα που προέκυψαν κατά το παρελθόν. Τα κράτη-μέλη είναι τα πρώτα που κρίνονται υπεύθυνα εάν ε, η διάσωση με τα ίδια μέσα δεν είναι αρκετή, δεν αρκεί. Πέρα από αυτό, όσον αφορά την έκθεση της Ελίζας και όσον αφορά και τις ε, τροπολογίες ε, που μάλλον θα προτείνουμε, θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, άρθρο 27 και άρθρο 30. Αυτά τα δύο άρθρα προσπαθούν να αποδυναμώσουν το ρόλο της Επιτροπής σε κάποιους τομείς. Και προφανώς αυτή είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, δηλαδή ο ρόλος της Επιτροπής σε όλο αυτό το θέμα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, βλέπουμε τις ε, διαπραγματεύσεις ε, που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις ενδεχομένως να βρεθούν κάποιες απαντήσεις για το θέμα της νομικής βάσης. Πάντως αυτή τη στιγμή με βάση το προτινόμενο άρθρο πιστεύουμε ότι πρέπει να εκχωρήσουμε στην Επιτροπή τις απαραίτητες αρμοδιότητες έτσι ώστε να μην αμφισβητείται η νομιμότητα όλης αυτής της διαδικασίας. Προφανώς ε, θα ήταν ε, καλύτερα για να αποφευθεί η σύγκρουση συμφερόντων ε, και να μην πολιτικοποιηθεί όλη αυτή η υπόθεση, να προβλέψουμε κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό μόρφωμα. Είχαμε ε, μία σχετική συζήτηση και όσον αφορά τον ε, ενιαίο μηχανισμό στήριξης, αλλά θεωρούμε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι ισχυρός για να καλύπτει τις νομικές της υποχρεώσεις. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις και πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πολύ σύντομα ε, θα μας εξηγήσει τι είναι δυνατό και τι όχι. Κατόπιν η Ελίζα προτείνει τις τροπολογίες 72 και 78 και εκεί αναφέρεται ένας όρος τα ε, δημόσια μέσα. Αυτό είναι ασαφές. Ε, οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης και ο προστατευτικός μηχανισμός, τουλάχιστον όσον αφορά το κοινό ταμείο εξυγίανσης, αυτά παραμένουν σε κρεμότητα. Και δεν ξέρω, ίσως, δεν ξέρω αν πρέπει αυτά να διευκρινιστούν σε αυτό τον κανονισμό. Ε, και μάλιστα φόσον πρόκειται για έναν όρο που δεν είναι ιδιαίτερα σαφής. Επίσης, ε, όσον αφορά την τροπολογία υπαριθμών 79, εκεί γίνεται λόγος για την απόλυτη προστασία των καταθετών. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι εξασφαλισμένοι οι καταθέτες και για να γίνει αυτό πρέπει να ψηφίσουμε για την έκθεση Σίμων που την περιμένουμε εδώ και δύο χρόνια. Αλλά τη στιγμή της ε, διάσωσης με τα ίδια μέσα είναι καλύτερα οι καταθέτες ε, να εντάσσονται σε αυτό το μηχανισμό πάνω βέβαια από τις 100.000 αντί να ξαναπληρώσουν οι φορολογούμενοι. Είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί όσον αφορά τις καταθέσεις, δηλαδή οι καταθέσεις ε, να μπουν απόλυτα ε, σε ένα σύστημα προστασίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ε, για τις πολύ μεγάλες καταθέσεις, τουλάχιστον κατά την άποψή μας. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω διευκρινήσεις για την τροπολογία υπεριθμών 34 που αφορά στη διαγραφή της υποχρέωσης να μετατραπεί το χρέος ε, κυρίως ε, όσον αφορά τις συμβατικές μεθόδους μετατροπής. Ίσως Ελίζα μπορείς να μας εξηγήσει λιγάκι ποιο είναι το ιστορικό αυτής της ε, τροπολογίας. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για την τροπολογία 65 και εκεί θέλουμε να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τι ε, κρύβεται πίσω από αυτή την τροπολογία που προβλέπει την διαγραφή της υποχρέωσης των κρατών μελών να ζητήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά αποφάσει που θα ε, συνεπάγονται δημοσιονομικές ε, υποχρεώσεις του κράτους μέλους. Όσον αφορά τώρα τις δικές μας τροπολογίες θέλω να υπογραμμίσω ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν πολλοί λόγοι το γιατί το σύστημα αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις τράπεζες και όχι μόνο για τις μεγαλύτερες. Διότι δεν μπορώ να καταλάβω ένα καθεστώς ε, το οποίο λέει μόνο οι τράπεζες υπό τον ενιαίο ποπτικό μηχανισμό θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα κοινό σύστημα εξυγίανσης, σε, ένα συγκεκριμένο ταμείο και υπό μια συγκεκριμένη αρχή, ενώ οι μικρές τράπεζες αφήνονται στη μοίρα των κρατών μελών. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι τα μικρά κράτη-μέλη τότε κάθε 20 χρόνια ε, θα ε, καταφεύγουν στο σύστημα εξυγίανσης των τραπεζών και αυτό για το οποίο πιέζει τώρα η γερμανική κυβέρνηση και είναι απομονωμένοι οι Γερμανοί με τη θέση τους αυτή στην Ευρωζώνη. Κατ' ουσίαν οι Γερμανοί προτείνουν οι οικονομίες που μοιάζουν λιγάκι με την οικονομία του μονάχου ε, θα πρέπει να έχουν το δικό του σύστημα τραπεζικής εξυγίανσης που σημαίνει ότι δεν έχουν την εμπειρία αυτές οι οικονομίες να αντιμετωπίζουν πραγματικές περιπτώσεις εξυγίανσης. Ε, γι' αυτό οι Ηνωμένες έχουν ένα ομοσπονδιακό σύστημα εξυγίανσης και ομοσπονδιακή αρχή εξυγίανσης. Έχουν ε, λόγο που το κάνουν αυτό γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει ε, ε, ένα εργαλείο χρηματοδότησης που θα εμποδίσει όλα αυτά να μετακυληθούν τελικά στους φορολογούμενους. ότι το τραπεζικό σύστημα κάποιων κρατών πολύ καλά και στη Γερμανία και στην Αυστρία ελοχεύει ο κίνδυνος και αυτό είναι εκείνο που οδηγεί τους Γερμανούς να εκφράζουν αυτή τη θέση. Ελοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος τα ε, θεσμικά συστήματα προστασίας αυτά ήδη κάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς και θέλουν τώρα να το περάσουν στους Ευρωπαίους. Και επειδή κάνουν αυτό το μεγάλο κομμάτι της δουλειάς, γι' αυτό δεν υποχρεούνται να πληρώσουν μεγάλα ποσά στις ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως ε, άλλες τράπεζες που είναι υποθεσμική προστασία. Και γι' αυτό τον λόγο αυτό όλο πρέπει να γίνει, αυτά που γίνονται στη Γερμανία να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκθεση Σίμων ε, ε, τα θεσμικά συστήματα προστασίας ε, θα τα προσιάσει ως ένα, μία από τις δυνατότητες για την προστασία των καταθετών και όσοι αυτοπροστατεύονται να πληρώνουν λιγότερα στο κοινό ταμείο εξυγίωνσης. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα και επιπλέον πρέπει να δούμε με απόλυτη σαφήνεια πώς μπορούμε να ζητάμε από τις τράπεζες να εξυγιανθούν υποχρεωτικά Όπως είπε η Σιλβί θα πρέπει να υπάρχουν ε, για τα κοινοβούλια ε, τα ίδια δικαιώματα ε, λογοδοσίας. Θα πρέπει να ζητάμε από τα κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρχει ίδια υποχρέωση λογοδοσίας και ενημέρωσης. Πιστεύουμε τελικά θα πρέπει να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι αυτοί οι δημόσιοι και ιδιωτικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης ε, ε, να αντικατασταθούν από το Ταμείο Εξυγίανσης. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω, να πω ότι στηρίζουμε τα περισσότερα από αυτά που προτείνει η Ελίζα, εκτός από τις ε, τροπολογίες που σας ανέφερα. Θα ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις, θα καλέσουμε όλους τους συναδέλφους να εργαστούν με ταχύ ρυθμό, γιατί η Κορίνα έχει δίκιο προηγείται πάντα η ποιότητα, αλλά εδώ νομίζω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένα από τους Ευρωπαίους και Μεταρρυθμιστές. Από την ΚΟΕ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ βέβαια δεν είμαι ο, ο ο συνάδελφος κόλλησε στη, στον δρόμο και δεν μπορεί να έρθει στο ταξίδι του, εν πάση περιπτώσει. Και δεν μπορέσαμε κάπως και να συμφωνήσουμε, αλλά η δική μου γνώμη είναι ότι σε γενικές γραμμές την έκθεση θεωρούμε σωστή, ε, ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα ε, που ε, εγώ τα θεωρώ ότι είναι προβλήματα, συγκεκριμένα το θέμα αυτού του περίφημου bail-in της διάσωσης με ίδια μέσα. Το όλο νόημα είναι να προστατεύσουμε τους φορολογούμενους. Από την άλλη όμως δεν είμαι απόλυτα σίγουρος κατά πόσο μπορούμε να τους προστατεύσουμε με τη διάσωση με ίδια μέσα. Αφενός πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό το κατόφλι ε, προστασίας των 100.000 παραμένει εξασφαλισμένο, δεν συζητάμε γι' αυτό, αλλά αυτοί που είναι πάνω από τις 100.000 που κατ' ουσίαν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές ε, μπορεί να χάσουν ένα μεγάλο κομμάτι κομμάτι της ε, περιουσίας της. Άρα δηλαδή ε, τελικά μήπως ε, με τον τρόπο αυτό θα ξαναδρομολογηθούν κρατικές ενισχύσεις για να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Αυτό μπορεί να ισχύει κυρίως για τις ασφάλειες και για τις συντάξεις γύρατος. Ε, εάν σε αυτές ισχύει το Μπελίν, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Και τίθεται και το ερώτημα, μήπως κατ' ουσίαν εδώ πρόκειται για την μετακύληση ε, ποσών και ευθυνών. Αυτό είναι το μόνο που με απασχολεί σε σχέση με το Μπελίν. Ε, κατά τα άλλα, ο κύριος Τόμας Χέντελ θα έρθει κάποια στιγμή στην επόμενη σύντηση και σίγουρα θα συμβάλλει πιο αποφασιστικά. Ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα στον κύριο κατάλογο. Ο κύριο Κλίν. Ευχαριστώ πολύ Σάρων. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά. Γι' αυτό εγώ θα κάνω μόνο λίγες ε, παρατηρήσεις. Να πω το εξή ότι αυτό το θέμα το βρίσκω πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο λυπάμαι πάρα πολύ ε, που όταν παρουσίασε την έκθεση η Ελίζα ε, ήταν παρόντες πολύ λίγοι συνάδελφοι. Πρέπει να προσέξουμε να μην πέσουμε στην παγίδα, να βρούμε λύσεις ε, για τον SRM που δεν θα καλύπτονται με όλα αυτά που αναφέρονται παραδείγματος σε σχέση με τον BRD. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω όπως και στην ΕΜΠΑ και στο SSM να Κάνουμε και εδώ το ίδιο, δηλαδή τους ε, σκιώδης ηγητές ε, κατά κάποιον τρόπο να τους βάλουμε να ε, συνεργαστούν και η ομάδα BBRD να συμπεριληφθεί στον SRM. Όσον αφορά τώρα το θέμα, πράγματι σωστά τα είπε η Κορίνα, μόνο που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να διασφαλίσουμε την ποιότητα. Συγκεκριμένα η ημερομηνία, η διορία που έχουμε για τις ε, τροπολογίες είναι πολύ γρήγορα ε, δημιουργεί πρόβλημα και το ότι δεν υπάρχει χρόνος νομίζω ότι αυτό είναι εις βάρος της ποιότητας. Όσον αφορά τώρα την έκταση, εγώ δεν συμφωνώ εδώ με τον Σβέν. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι έχει νόημα να διαμορφώσουμε την εποπτεία διαφορετικά από το μηχανισμό SRM ή αντίστροφα αν θέλετε. Δηλαδή αν συμπεριλάβουμε όλες τις τράπεζες, ακόμα και τα μικρά ταμιευτήρια, τότε κατά την άποψή μου όχι μόνο ε, προσκρούμε στην αρχή της ε, επικουρικότητας, στην αρχή της ε, ενιαίας διαμορφώσης αλλά και της επικουρικότητας. Επίσης, Βεν, αν κάνουμε αυτό που είπες εσύ, τότε αυτό θα σημαίνει ότι ε, αρχίζει πλέον να μην ισχύει η αρχή της ε, κοινή εποπτείας και γι' αυτό δεν το θεωρώ αυτό ε, ιδιαίτερα λογικό. Όσον αφορά τώρα τους μηχανισμούς εξυγίανσης εδώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εξή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Αρχές Εποπτείας παρακολουθούν την κατάσταση και εκείνες αποφαίνονται κατά πόσον μία τράπεζα ε, είναι βιώσιμη ή όχι. Αλλά ε, το Ταμείο Εξυγείωσης και η Επιτροπή λαμβάνουν την τελική απόφαση. Κατά πόσον αυτός είναι ο σωστός δρόμος, νομίζω αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, να δούμε μήπως τελικά αυτή είναι μία πολύ περίπτωση περίπλοκη διαδικασία και θέλω να κάνω και το εξή ερώτημα. Εδώ νομιμοποιείται η Κομισιόν ως, ε, να εμφανίζεται ως ο καθοριστικός παίκτη. Νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα ξανασκεφτούμε. Όσον αφορά τώρα το Ταμείο. Γνωρίζουμε βέβαια όλοι μας ότι πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο και γνωρίζουμε ότι το ταμείο δεν μπορεί να πρικοδοτηθεί μια νυχτή. Χρειάζονται πολλά χρόνια, ίσως ούτε καν τα 10, ίσως και 15 χρόνια μέχρι να έχουν μπει όλοι στο ταμείο αυτό και έτσι πράγματι να μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ισχυρό, δυνατό ταμείο. Νομίζω ότι τώρα γίνεται λόγος για 45 δις ε, πρέπει να σας πω ότι για την Ευρωζώνη αυτό δεν αρκεί, πολύ μικρό το ποσό. Στη Γερμανία ε, το ταμείο που έχει ήδη αποφασιστεί και λειτουργεί ήδη έχει ως ε, στόχο πρικοδότησης μόνο του 70 δις. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν ταιριάζουν και το ότι όσο το Ταμείο αυτό δεν είναι απόλυτα πρικοδοτημένο ότι χρειάζεται ε, οικονομική προστασία, backstop, αυτό είναι σαφές. Μόνο που ποιος θα το κάνει αυτό, αυτό δεν είναι σαφές. Και οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί κατά την άποψή μου δεν είναι επικοδομητικές, διότι απλά με παρακάμψεις απλά φτάνουν και πάλι ε, στον φορολογούμενο. Είτε είναι το SRM, είτε μια άμεση αναχρηματοδότηση στην αγορά από το Ταμείο. Σε τελική ανάλυση όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο εφόσον υπάρχουν εγγύησεις και οι εγγύησεις ε, προφανώς ε, φτάνουν ε, στον φορολογούμενο. Όσον αφορά τη χρήση του Ταμείου και την απόφαση που θα ληφθεί, όλα αυτά πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αναφέρεται να αποφασίσουν έξι και δύο εξ αυτών ανήκουν ε, στα κράτη-μέλη, στα μέλη, στα κράτη-μέλη. 17 είναι αυτή τη στιγμή. Προστίθεται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή από τις 6 οι 2 εκπροσωπούν τα 18 κράτη-μέλη. Αυτό κατά την άποψή μου ε, δεν είναι ισορροπημένο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και τα πολύ μικρά, με ίσο βάρος ψήφου. Και εδώ για 18 κράτη έχουμε μόνο δύο ε, που μπορούν να ψηφίσουν και η ψήφος τους είναι η όπως αυτή της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό που επίσης πρέπει να διευκρινιστεί είναι τι γίνεται με τα εθνικά ταμεία που είναι εν τη γενέση τους έχουμε στην ε, Γερμανία, στην Αυστρία, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά τα εθνικά ταμεία αυτή τη στιγμή ε, χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες όμως με διαφορετικά κριτήρια και ο στόχος είναι επίσης διαφορετικός. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται θα αντιοχητευτούν και για διαφορετικούς σκοπούς και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη των χρηματοδοτήσεων από τα χρηματοδοτικά Ινστιτούτα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται τα εθνικά αυτά ταμεία και παράλληλα θα αρχίσει να χρηματοδοτείται και το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Ε, νομίζω σιγά σιγά αυτό θα καταλήξει σε μια ε, χρηματοδοτική επιβάρυνση που είναι υπερβολική. Κατά τα άλλα, το ερώτημα πού θα εγκατασταθεί το Ταμείο. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ας είναι εδώ στις Βρυξέλλες ε, το ταμείο αυτό. Ε, κατά τα άλλα, όπως είπε και η Κορίνα, υπάρχει και η δεύτερη, ο δεύτερος πολύ σημαντικός πυλώνας της ε, Τραπεζικής Ένωσης και δεν πρέπει να την σπάσουμε την Τραπεζική Ένωση. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουμε την εποπτεία στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο νέος μηχανισμός εξυγίανσης, το SRM, δεν θα είναι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, την Κεντρική, αλλά θα έχει έδρες Βρυξέλλες. Δεν ξέρω, δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι δυσχεραίνει την κατάσταση και τουλάχιστον ας το σκεφτούμε. Και κάτι άλλο, ένα τελευταίο σημείο. Λέμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται στο άρθρο 114 TFUE πρόκειται για ένα μέτρο ε, με στόχο την ενίσχυση της κοινή αγοράς. Γι' αυτό και γίνεται επίκληση αυτού του άρθρου. Αν όμως είμαστε ειλικρινείς, κατ' ουσίαν πρόκειται για ενίσχυση μόνο ενός τμήματος της κοινή αγοράς, της ευρωζώνης δηλαδή. Και αν θέλετε, de facto, ε, πρόκειται για ε, δυσχερέστερη κατάσταση στην οποία θα βρεθεί η κοινή αγορά των 28. Ε, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θα υπάρξει ένας κανονισμός, αλλά στην BRD λέμε ότι αυτό δεν φτάνει πρέπει να υπάρξει μια οδηγία που δεν θα είναι τόσο αυστηρή. Εγώ δεν είμαι νομομαθής ούτε νομικός, αλλά διερωτώ με μήπως ε, εδώ κάποιος ε, τα ερμηνεύει πάρα πολύ ευέλικτα. Ίσως λοιπόν θα ήρθε νόημα να επιληφθούν το θέματος οι νομικοί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σάρων. Εγώ θα ήθελα σύντομα να τονίσω καταρχήν τη σημασία του θέματος που συζητάμε σήμερα, το πώς ε, συνδέεται με την Τραπεζική Ένωση και το γεγονός ε, ότι θα, όταν θα ολοκληρώσουμε όλο αυτό το οικοδόμημα, τότε μπορεί αυτό να επιφέρει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα και μείωση του κόστους ε, του δανεισμού στα διάφορα και το ίδιο ισχύει και στις διασυλλογικές ε, συναλλαγές και χρηματοδοτήσεις γιατί πολλές ε, φορές έχουμε πολύ μεγάλο κόστος για να δανειστεί μια επιχείρηση από μια άλλο χώρα. Αυτές τις τελευταίες εβδομάδες ε, πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό και εγώ θέλω να τονίσω τέσσερα θέματα που θεωρώ ιδιαίτερα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Καταρχήν, το θέμα του να υπάρχει ένας μηχανισμός οικονομικής στήριξης, ένα backstop ε, θα είναι ένας μηχανισμός δανεισμού που θα μπορεί να επιφέρει ε, την εμπιστοσύνη στο σύστημα και γι' αυτό θα πρέπει ήδη να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε ότι αυτό το backstop να μπορεί να είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός που θα είναι αντικείμενο διαχείρισης με κοινοτικού κανόνες και με κανόνες ευρωπαϊκής προέλευσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αρχίσουμε να δίνουμε ένα μήνυμα εμπιστοσύνη στους πολίτες και στους καταθέτες. Δεύτερον, θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα προσφυγής ε, των αποφάσεων, των αποφάσεων του Συμβουλίου. Πολλές από αυτές θα είναι ε, αποφάσεις που θα έχουν σε ισχύ αφού θα έχουν ε, εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να εκτελεστούν γρήγορα αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών. Δεν έχει αναφερθεί ιδιαίτερα αυτό το σημείο, αλλά εγώ θα ήθελα να το επισημάνω. Τρίτον, ο τρόπος ε, που ένας, ε, μια ευρωπαϊκή οντότητα εξυγένσης θα σχετιστεί με τις εθνικές οντότητες. Αυτό επίσης είναι ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω. Και τέλος, ποιος είναι ο τρόπος συσχέτιση σχέσεων μεταξύ Κομισιών και του Συμβουλίου. Δηλαδή θα λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις από το Συμβούλιο και κατόπιν θα δίνεται μία συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτά θα επικεντρωθούν οι τροπολογίες που θα παρουσιάσω και εγώ θέλω να πω ότι ελπίζω να μπορέσει να στεφθεί με επιτυχία αυτό το έργο και Είναι προφανές ότι θα στεφθεί με επιτυχία γιατί θέλουμε να ελπίζουμε ότι μέχρι να φτάσουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές ε, θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ο συνάδελφος Βόλφ Κλίντς είπε πολλά από αυτά που ήθελα να πω και εγώ. Ε, θέλω να αφαιρθώ λιγάκι στον τρόπο χειρισμού των μικρών τραπεζών. Ε, θέλω να σας πω ότι δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Σβεν Γκίγκολτ, δηλαδή ότι... Ε, οι συνεταιρισμοί τραπεζών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν θα είναι σε θέση να προβούν σε εξυγίανση απλά και μόνο ε, διότι υποτίθεται δεν τις αφορά. Κάθε άλλο, η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο. Η πραγματικότητα δείχνει ότι τέτοιου είδου ε, μία πολλές φορές ε, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και μάλιστα να τις αντιμετωπίσουν, να τις εξηγιάνουν με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Νομίζω λοιπόν, όπως είπαν και πολλοί προλαλήσαντες, ε, θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά με ποιο τρόπο θα ε, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις μικρές και τις μεσαίες τράπεζες σε, αυτόν, σε αυτό το ταμείο. Στη, με την κρίση αποδείχτηκαν κάποιες ε, επιτυχημένες εξελίξεις και αυτές να παραμείνουν. Και εδώ εννοώ τράπεζες που θα πρέπει να υπολογιστεί το τι θα καταβάλουν στο ταμείο. Βέβαια, εάν ένα ταμείο καλύπτει πλήρως ε, τους κινδύνους, τότε πρέπει να διερωτηθούμε τι θα καταβάλουν οι τράπεζες αυτές, αλλά και στην περίπτωση αυτή τι να το κάνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο, τι το χρειάζονται. Είτε λοιπόν το εξή δεύτερο ερώτημα. Έχει νόημα το Ταμείο να επεκτείνεται και σε αυτές τις τράπεζες. Ε, θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες λύσεις έτσι ώστε και αυτές οι τράπεζες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτά ε, τα οποία συζητάμε κοστίζουν χρήματα. Τα χρήματα που θα καταβάλουν οι τράπεζες ταμείο έρχονται από τον πελάτη, από πού αλλού να έρθουν. Είναι λοιπόν απολύτως ε, απαραίτητο να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση των τραπεζών και να μην αφήσουμε ε, κάποια Ινστιτούτα που έχουν δημιουργήσει ολόκληρα συστήματα να επιβαρύνονται διπλά, απλά και μόνο διότι ήταν πολύ πιο συνετά και φρόνημα από άλλα. Ο κύριος Χοκμάγκ έχει το λόγο, Γκούνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν εδώ είναι πολύ πεπισμένος ότι αφού άκουσα όλους τους συναδέλφους εδώ και τις σκέψεις τους για το τι να κάνουμε με την εξυγίανση και την ανάκαμψη των τραπεζών, ότι είναι πολύ σημαντικό να τεθεί σε εφαρμογή οδηγία το συντομότερο, αλλά και ως βάση για αυτή την νομοθεσία γιατί διαφορετικά βλέπω να υπάρχει προφανής κινδυνός ότι οι διάφορες φιλοσοφίες για την επίλυση των προβλημάτων ε, θα καταστήσουν αμφίσιμες αυτές τις οδηγίες. Αν ε, δεν έχουμε συνεκτικότητα θα δημιουργηθεί έλλειψη διαφάνειας αλλά και δυνατότητα κακοπραξίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ζωτικό όπως ε, και να συνάδει αυτό το νομοθέτημα με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Τώρα ε, υπάρχουν πάρα πολλές ενσορπίες και πρέπει να ρυθμίσουμε την ε, νομοθεσία για το σύστημα των καταθέσεων και κατόπιν να προχωρήσουμε. Η Κομισιόν πρότεινε την πρόταση για τον SRM βάσει του κειμένου για την ε, ανάκαμψη. Όμως αυτό υπογραμμίζει ότι πρέπει να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά τα θέματα και να τα διορθώσουμε και να κάνουμε τα βήματα με μια λογική σειρά. Κάτι ακόμη που νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε έχει να κάνει με τα όσα είπα. Είναι η διαδικασία της διάσωσης με ίδια μέσα που πρέπει να είναι η ίδια Ό,τι και κάνουμε, δεν μπορούμε να έχουμε έναν τρόπο διάσωση με ίδια μέσα και να έχουμε, δηλαδή να ρυθμίσει το μηχανισμό SRM και άλλο τρόπο διάσωση με ίδια μέσα ε, ε, στην ε, νομοθεσία περί εξυγίανσης. Έτσι λοιπόν αυτό τονίζει τι γίνεται και πόσο προβληματικό είναι να έχουμε παράλληλα δύο νομοθετήματα. Και κάτι ακόμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτό έχει συνέπειες ε, για τη συζήτηση για τον SRM. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να θεσπίσουμε ένα σύστημα όπου οι τράπεζες είναι στο δυνατόν πιο εύρωστες, πιο υγιείς και όλοι όσοι χρηματοδοτούν ή επενδύουν είναι διοκτήτες τράπεζες να ξέρουν ότι δεν θα μπορούν να αποφύγουν τις απώλειες ή τις προκλήσεις των απολειών. Αλλά ταυτόχρονα εγώ νομίζω ότι αυτό και υπογραμμίζει την ανάγκη για σταθερότητα και την αναγκαιότητα κυβερνήσεις σε καιρό κρίσης να διασφαλίσουν τη σταθερότητα να άκουσα τη συζήτηση για τα backstop στους μηχανισμούς χρηματοοικονομικής στήριξης. Ξέρω ότι όλοι θέλουν να υπάρχει αντιστοιχείος μηχανισμός κάπου, αλλά όχι στην ίδια την αυλή. Το backstop ε, είναι προτιμητέο να βρίσκεται κάπου αλλού και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα σε ποιε επιθέσεις, γιατί αν δημιουργούμε ένα σύστημα όπου κυβερνήσει και τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση ή μπορούν να αποφύγουν την ευθύνη που έρχεται από το γεγονό ότι έχουν μια ευκαιρία να αναλάβουν δράση, τότε θα υπάρχει πάντοτε ελπίδα ότι κάποιος άλλος θα το λύσει το πρόβλημα. Και ακούσαμε όλοι τη συζήτηση για το Ταμείο Εξυγίανσης και νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ε, όσο μεγάλο και είναι το Ταμείο Εξυγίανσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάλι δεν θα αρκεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις αν έχουμε μια ευρύτερη συστημική κρίση. Και αν δεν έχουμε την ευκαιρία να δράσουμε με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία, ο κίνδυνος είναι ότι όλοι θελπίζουμε ότι κάποιοι άλλοι θα λύσουν το πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα θα το συναντήσουμε όταν θα φτάσουμε σε στάδιο ολοκλήρωση αυτής της νομοθεσίας, αλλά πρέπει να αποσαφινιστεί. Μάλιστα, ευχαριστώ. Και εγώ έχω βάλει τον εαυτό μου στον κατάλογο των ομιλητών. Καταρχήν, ε, με αυτή την πρόταση αντιμετωπίζω διάφορα προβλήματα, γιατί αφενός πολιτικά συμφωνώ απόλυτα με τη σημασία να συσταθεί αυτός ο μηχανισμός και να ενδυναμωθεί το όλο project της Τραπεζικής Ένωσης. Αλλά όσο κοιτάζω αυτό το νομοθέτημα, τόσο περισσότερο Αναρωτιέμαι ε, αν ε, όλα αυτά θα έπρεπε να είναι σαν νομοθετήμα γιατί έρχεσαι να μοιάζει πολύπλοκο. Συμφωνώ όμω, είπε ο Γκούναρ ότι το βασικό έγγραφο που έχει να κάνει με τον Μπέιλιν και όλου του κανόνες και με το η ευελιξία υπάρχει ή όχι υπάρχει στην οδηγία για την ανακάμψη και την εξυγίανση και δεν μπορούμε να έχουμε ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει διαφορετικά πράγματα στο θέμα της εξηγήσεως των τραπεζών. Θα ήταν ιδιαίτερα ατυχές αν επειδή κάποιος ε, είναι στον νέο εποπτικό μηχανισμό τελικά κατέληγε σε χειρότερη κατάσταση λόγω του πώ έχουν εισαχθεί κάποια στοιχεία σε έναν κανονισμό και πώ συνδυάζονται με άλλα. Φυσικά χρειάζεται να υπάρχει κανονισμό για να συσταθεί η αρχή τη εξυγίαση. Και φυσικά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν μια οδηγία. Όμως, εγώ θεωρώ ότι πρέπει στο μέτρο του δυνατού να μην ε, κάνουμε απλώς ε, παραθέσεις, αλλά να έχουμε παραπομπές κατευθείαν στην ομοθέσια, Στην BRRD έχουμε ένα θέμα για το ποιος θα πυροδοτεί την εξυγίανση και φυσικά αυτό αντικατοπτρίζει εδώ και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Κομισιόν. Έχει υποθεί συχνά ότι η αρχή της εξυγίανσης που προτείνουμε εδώ κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ένα παράλληλο μηχανισμό με το FDIC των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά με κανένα τρόπο δεν μπορούν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών να λειτουργήσουν όπως λειτουργούν η πάλι του FDIC δεν πρόκειται εκεί για ένα μηχανισμό εξυγίανση μόνο, αλλά έχει όλη την εμπειρογνωμοσύνη και για την χρηματοοικονομική εποπτεία. που χρειάζεται όταν μιλάμε για εξυγίανση τραπεζών. Όταν μιλάμε για κάποιο μεγάλο ίδρυμα, ακόμη και στις Ηνωμένε Πολιτείες, γίνεται έρευνα για να δουν τι άλλο πρέπει να κάνουν. Και νομίζω ότι πρέπει όταν ε, μιλάμε και για θέματα έδρας πρέπει να το δούμε αυτό και πώς πρόκειται να λειτουργήσει ο μηχανισμός εξυγίανσης. Η όλη ιδέα είναι ότι ε, θα έχουμε τους ε, κανόνες του κράτους μέλους υποδοχής που θα ισχύουν και αυτό θα το δεχτεί το κράτος μέλος που φιλοξενείται. και ε, αν ε, δεν είναι προετοιμασμένο το κράτος μέλος ε, που φιλοξενείται να κάνει να οπισθοχωρήσει, τότε πηγαίνουμε στο πολλαπλό σημείο εισόδου. Και πιθανόν θα έχουμε διεθνείς συμφωνίες, όπου θα μπορούμε να έχουμε ένα ενιαίο σημείο εισόδου. Αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία υπαναχώρησης. αν τελικά υπάρχει υπερβολική παρέμβαση από το άλλο κράτος μέλος. Αν όμως το δει το θέμα κανείς απ' έξω, εμένα είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Η όλη δομή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει δυνατότητα opt-in-out, αλλά επίσης ε, ε, εφαρμόζεται και σε σύνολα τραπεζών που καθορίζονται από διάφορα κριτήρια. Φυσικά όλες οι τράπεζες είναι στον ε, νέο μηχανισμό. Εγώ θεωρώ ότι το να λέμε ότι κάποιοι μόνο θα υποβάλλονται, κάποιες μόνο τράπεζες θα υποβάλλονται σε αυτό, είναι κάπως ε, προβληματικό. Γιατί ουσιαστικά υποσκάπτεται εδώ η ιδέα του να έχουμε ενιαίους κανόνες. Και νομίζω ότι τελικά μπορεί να το μετανιώσουμε αυτό. Ίσως ο καλύτερος τρόπος να το μετωπίσουμε είναι να έχουμε μια ρήτρα αναθεώρηση που να λέει ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί αυτό το υποσύνολο. Εγώ δεν είμαι καν πεπισμένη ότι θα γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον και αν πρέπει να περιοριστούμε εδώ ε, στον SSM. Αυτό θα εξαρτηθεί από το μηχανισμό, από τον backstop που θα τεθεί σε λειτουργία. Ξέρω ότι υπάρχει ευαισθησία σε κάποια κρατημέλη. Μπορεί να μην ήθελαν να ενταχθούν στο σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρήση του ταμείου, έχω μπερδευτεί. Φαίνεται ότι έχουν πάρει κάποια στοιχεία εξυγίνησης από την BRRD και λέει ότι δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε κρατική ενίσχυση. Όμως ε, κανένα τέτοιο σχέδιο εξήγησης τραπεζών θα πρέπει να κάνει αναφορά στο ταμείο. Αυτό δεν αποτελεί τμήμα του σχεδίου εξηγήσης, αλλά θα χρησιμοποιείται ως κονδύλι έκτακτης ανάγκης. και θα πρέπει να καλύπτεται το κόστος της εξυγένσης ε, αντί της χρεοκοπίας και να γίνεται κάποιες επιλογές αν θα ε, διασωθούν κάποιες μικρές και μεσές επιχειρήσεις ή κάποιες κατηγορίες καταθετών. Όμως ε, κάποιοι άλλοι μπορεί τους χάρη να πάνε σε χρεοκοπία. Έτσι λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμείο. παραδείγματο χάρη να σταματήσει μια κατάσταση που μπορεί να μα κοστίσει τέσσερις φορές παραπάνω. Αυτή θα είναι η πρωταρχική στόχη του Ταμείου. Αρχίσαμε να συζητάμε ότι θα αποτελεί ένα είδο backstop, αλλά αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις κοινωνικέ του υπηρεσίες για την τράπεζα, ε, τότε θεωρούμε ότι όλο ο ενιαίο μηχανισμό εποπτεία είναι πολύ μεγάλο για να αποτύχει και ότι τελικά θα τα διασώσουμε ό,τι και να γίνει. Πρέπει και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά που λέμε. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι η παρέμβαση του Ταμείου είναι, γίνεται σε έσχατη, ως έσχατη λύση. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θα ισχύει στα κράτη-μέλη. Γιατί δεν μπορούμε, παραδείγματο χάρη, να έχουμε την περίπτωση που η Σουηδία θα έχει ένα ταμείο που το έχει συστήσει από εισφορά τράπεζα και θα μπορεί να υποβάλλεται σε κανόνε κρατική βοήθεια, αλλά δύο άλλε χώρε θα κάνουν ένα κλαμπ ε, που δεν θα σέβεται αυτού του κανόνε κρατικών ενισχύσεων. Θα πρέπει όλα να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί να υπάρχει ειδικό καθεστώ. Και άλλα έχω να πω. Έχω και άλλα αλλά μάλλον θα καταθέσω τροπολογίες σχετικά. Αν το Ταμείο τελικά τεθεί σε λειτουργία και κάνει πράγματα, τότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά έχει αξία. Δηλαδή, αν θα δίνουν εισφορές στα ιδιωτικά ιδρύματα και κατόπιν χρησιμοποιούμε τα χρήματα, πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι έλεγχοι ex για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα όπως πρέπει. Έχει να κάνει με κανόνες οικιακής οικονομίας. Δεν θα κυνηγάμε μάγισσες, δεν πρόκειται και κυνήγι μαγισσών. Αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί μπορεί να υποσχεζόμαστε ότι την πρώτη φορά δεν θα πάνε καλά τα πράγματα και θα μάθουμε μέσω της εμπειρία. Και αν δεν γίνονται τέτοιε αξιολογήσει, τότε δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση και ούτε θα τα καταφέρουμε τη δεύτερη ή την τρίτη φορά. Θα προσπαθήσω λοιπόν ε, να καθέσω κάποιες τροπολογίες σχετικές με το όσα είπα. Έχουμε και κάποιους άλλους στον κατάλογο. Θα το διαβάσω γιατί μπορεί να αναρωτιέστε πότε θα έχετε το λόγο. Αυτή ήταν η σειρά. Όχι εσείς ακόμη. Είστε τελευταίος. Η Άστριτ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη μου έλευση. Ήμουν σε άλλη συνεδρίαση στη γυναικών για τις ποσοστώσεις συζητούσαμε και γι' αυτό δεν μπόρεσα να έρθω από την αρχή. Λοιπόν, Θα πω μερικά γενικά. Και να τονίσω τη σημασία του κανονισμού αυτού που αφορά ένα τόσο σημαντικό θέμα και με τόσο σοβαρές επιπτώσεις. Γιατί η δημιουργία ενός τρικτικού μηχανισμού, ενιαίου μάλιστα, είναι κατ' αναγκαία. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω πρέπει να επιδείξουμε επιμονή μπροστά στις προσπάθειες που γίνονται να αποδομηθεί η πρόταση αυτή εκ μέρους ορισμένων κυβερνήσεων που γνωρίζουμε όλοι και του Συμβουλίου. Εγώ πιστεύω ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ σωστά έπραξε με την πρότασή του που είναι σοβαρή παρά το νομικό της υπόβαθρο που είναι κάπως αδύνατο. Υπό τη συγκυρία αυτή βέβαια πιστεύω και εγώ όπως και εκείνος ότι έτσι έπρεπε να γίνει διότι η στήριξη μιας τράπεζας παραμένει κάτι πολύ λεπτό και δύσκολο και μπορεί να σημαίνει και αποτυχία κατάλληλης εποπτείας λόγω όλων όσων σημαίνει. Πρέπει να είναι τα πράγματα να γίνουν σαφή χωρίς ζώνες σκιάς. Νομίζω ότι η ανεξαρτησία των αρχών που θα δημιουργήσουμε είναι το κλειδί για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα διότι θα χρειαστεί να πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι αποφάσεις των αρχών αυτών να λαμβάνονται όχι με βάση εθνικά συμφέροντα αλλά με βάση το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Ό,τι θα επέτρεπε στα κράτη-μέλη να να επαναπροσανατολιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση, θα ήταν θετικό και το αντίθετο αρνητικό. Αυτό αφορά και τη δομή της λήψης αποφάσεων, τον μηχανισμό την κατανομή των εξουσιών home και host όλα αυτά είναι λεπτά επαναλαμβάνω λοιπόν ότι νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή για όλα αυτά τα θέματα γιατί πιστεύω ότι τα κράτη θα θελήσουν να ξαναπάρουν από τη μία αυτό που αφήνουν απ' την άλλη. Να το προσέξουμε αυτό και η Κομισιόν είμαι βέβαιη ότι θα φανεί πολύτιμο σύμμαχος για μας εάν πράγματι συμφωνήσουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης νομίζω είναι ίσως νωρίς να μιλήσουμε για τροπολογίες θα καταθέσω αλλά δεν θα τα αναφέρω τώρα. Επί των αρχών νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε ένα μηχανισμό, ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης ως βασικό θεμέλιο για την, για την Τραπεζική Ένωση. Αλλά να μην οικοδομήσουμε ένα κάτι που δεν θα στέκει στα πόδια του σταθερά και τελικά καταλήξουμε να έχουμε περισσότερα προβλήματα από τη λύσεις. Αυτό ήθελα να σας πω σήμερα. Και ίσως θα επανέλθω στις τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Μερικοί ζητάνε δύο φορές το λόγο, δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό. Γιατί έχουμε στο τέλος και ψηφοφορία. Και είναι πολλοί ομιλητές. Ο Πέτρος Σίμων. Ευχαριστώ πολύ Σάρον. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάτι που είπε προηγουμένως ο Γκούνο Χακμακ ε, και το είπε και ο Αυστριακός συνάδελφος. Συγκεκριμένα στο ποιες τράπεζες ε, στο μέλλον ε, θα λαμβάνονται υπόψη και το θέμα που είπε και ο κύριος Χοκμαρκ, ε, δηλαδή το θέμα της ταύτισης με την Τραπεζική Ένωση. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι έχουμε Τραπεζική Ένωση αλλά προχωράμε με τελείω διαφορετικές ταχύτητες. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε έτσι ώστε στο τέλος όλα αυτά κάπως να ταιριάζουν. Και συμφωνώ με τον Γκούναρ πρέπει ε, να είμαστε προσεκτικοί, ε, την εποπτεία τη ρυθμίσαμε, αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι και την νομοθεσία για τη διάσωση ε, και την ανάκαμψη και για την εγγύηση των καταθετών έτσι ώστε να έχουμε ένα κοινό ε, πεδίο, θεμέλια και μετά να προχωράμε πάνω σε αυτά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο στόχος, ότι ναι μεν έχουμε το στόχο σε αυτά τα τρία θέματα αλλά όσον αφορά λεπτομέρειες και μεμονωμένα υποθέματα Εκεί πιέζουμε χωρίς όμως να γνωρίζουμε κατά πόσον υπάρχει ταύτιση των μεμονωμένων θεμάτων και μπορεί να προκύψουν μεγάλα προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν με απόλυτη σαφήνεια να αναφερθώ στο εξής. Εάν θεωρήσουμε στο θέμα της ευθύνης ότι πρέπει να υπάρχει κοινό κοινή ρύθμιση για ευθύνες και εγγύησεις θα πρέπει αυτομάτως να πούμε ότι μόνο ορισμένες τράπεζες θα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία. Και κατόπιν τούτου, όσον αφορά το επίπεδο, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον στην ευθύνη ισχύει το ίδιο επίπεδο όπως και στην εξυγίανση. Νομίζω λοιπόν εδώ πρέπει να προτείνουμε ακριβώς το ίδιο όσον αφορά και την εξυγίανση, δηλαδή αν θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και εδώ θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε το θέμα της εποπτείας. Και για να είμαι απόλυτα σαφής και εγώ πιστεύω ότι όσον αφορά τα θέματα που συζητάμε εδώ, Προφανώς και συζητάμε για ε, διασυνοριακές ε, τραπεζικές συνεργασίες. Δεν μιλάμε εδώ ε, για μικρομεσαίες ε, τράπεζες, κυρίως αναφορά τις ε, μικρές τράπεζες που πράγματι όλα αυτά χρήζουν ρυθμίσεων, μπορεί να υπάρξει κάποια απόφαση που να λέμε δεν θέλουμε αυτές να τις διασώσουμε, ας πτωχεύσουν αυτές οι μικρές και ας πληρώσουν οι καταθέτες. Αυτή όμως η απόφαση, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρχει, να είναι δυνατό να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα κάτι άλλο που ετέθη προηγουμένως, δηλαδή σε τελική ανάλυση ποιος είναι εκείνος που θα πυροδοτήσει την εξυγίανση, εδώ θέλω να αφαιρθώ σε αυτά που είπε η συνάδελφος κυρία Λούλινγκ, η οποία είπε στο μέλλον η αποτυχία μιας τράπεζας θα ισούται με την αποτυχία της εποπτείας. Σωστά και πρέπει να προσέξουμε, να δούμε μετά τι γίνεται με την εξυγίανση. Γιατί γίνεται συζήτηση πώς θα γίνεται εξυγίανση, θα γίνεται από μια επιτροπή. Κάποιοι άλλοι λένε να δούμε κατά πόσον εξυγίανση θα γίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ τώρα έχω πρόβλημα να τα καταλάβω όλα αυτά ε, και θα ήθελα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Γιατί μπορεί πράγματι να συμβεί η περίπτωση εκείνη όπου η αρχή η οποία είναι αρμόδια για να αποφασίσει για την αξυγίανση, η αρχή αυτή θα το αποφασίσει εν πάση περιπτώσει και το κράτος στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη τράπεζα, το κράτος να πει ακριβώς το αντίθετο, για χι λόγους, χι ψι Τότε το κράτος αυτό θα πρέπει να αγωνιστεί έτσι ώστε να μην υπάρξει, να μην τρομολογηθεί η εξυγίανση. Μπορείτε να φανταστείτε η Γερμανία να αρχίσει να πυροβολεί κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί δεν επιθυμεί να έχει μια συγκεκριμένη εξυγίανση. Καταλαβαίνετε ε, το κύρος, πόσο θα ε, τρωθεί το κύρος της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι είναι δύσκολα θέματα αυτά που πρέπει να τα συζητήσουμε, ίσως όχι σήμερα, αλλά επειδή μέχρι την Παρασκευή είναι η διορία, εντάξει θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή και όταν θα έχουμε δεσμευτικούς κανόνες να δούμε και το πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε την νομοθεσία και για τους τρεις τομείς. Okay, uh, thank you. Marianne. Η Marianne. Ευχαριστώ. εγώ κατάλαβα ότι εμείς ε, θέλουμε μια εσωτερική αγορά για τα 28 κρατημέλη και οι μηχανισμοί που θέλουμε να δημιουργήσουμε πρέπει να είναι ομοιόμορφοι. Έτσι οικοδομήθηκε και ο SSM. Αν δούμε στη συνέχεια ποιος ε, συμμετέχει στον μηχανισμό εποπτείας, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες ε, τράπεζες εντάσσονται σε αυτά τα συστήματα. Θα πρέπει να κάνουμε ένα παράλληλο με το μηχανισμό εποπτείας και να ε, συμπεριλαμβάνονται εδώ οι τράπεζες μόνο που είναι υπό την εποπτεία της ΕΚΤ. Όμως δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πάντοτε πίστευα ότι ο νέος εποπτικός μηχανισμός είχε επιλεχθεί ακριβώς επειδή θα έπρεπε να λειτουργεί το σύστημα με ένα οργανωμένο τρόπο και κατόπιν ε, κάναμε μια διάκριση για τις τράπεζες που ελέγχονται απευθείας από την ΕΚΤ και τις άλλες που σε πρώτο στάδιο βρίσκονται από τον έλεγχο μιας εθνικής αρχής σε πρώτο στάδιο, αλλά κατόπιν ε, εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου της ΕΚΤ και υπό αυτή την έννοια μπορεί πάντοτε να μιλάμε για μια τράπεζα που μπαίνει στο σύστημα ή αν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις μπορεί να ζητήσει από την ΕΚΤΕ να ελέγξει το Ίδρυμα αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα με το θέμα της εξυγίανσης των τραπεζών θα πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ των τραπεζών και μάλιστα εμείς αυτή τη διάκριση την κάναμε εδώ με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί. Και εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν εδώ και 6.000 τράπεζες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Γιατί αν ε, εισαγάγουμε διακρίσεις τότε το τοπίο θα είναι εντελώς πολύπλοκο και δεν θα έχουμε τα πλεονεκτήματα που θέλουμε. Διαφοροποίηση, ναι, διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την εισφορά των διάφορων τραπεζών στο ταμείο αυτό. Ναι, ανάλογα με το επιχειρηματικό τους μοντέλο, με την έκθεσή τους στον κίνδυνο. Ναι, εδώ μπορούμε να έχουμε μια διάκριση σε ό,τι αφορά την εισφορά των τραπεζών στο ταμείο, αλλά όχι διαφορετικού είδου διάκριση. Εγώ νομίζω ότι θέλουμε παραλληλισμό εδώ με τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό και πρέπει να μιλάμε ακριβώ για τι ίδιε οντότητε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας θυμίσω κάτι που έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος θα συμμετέχει σε αυτόν τον ενιαίο μηχανισμό. Σας υπενθυμίζω ότι αν μερικές χώρες εκτός Ευρωζώνης γίνουν, μπουν σε αυτό το ταμείο, τότε θα πρέπει να συμμετέχουν και στους υπόλοιπους μηχανισμούς, στην Ευρωζώνη δηλαδή. Αλλά θα διατηρηθεί έτσι η ακαιρεότητα της ενίας αγοράς. Εγώ εκπροσωπώ την Μπολονία και η χώρα αυτή είναι ακόμη έξω από την Ευρωζώνη αυτό το βήμα της Κομισιόν είναι η παναχώρηση σε σύγκριση με αυτά που είχαμε διαπραγματευτεί ως συμβιβαστικές προτάσεις για τον εποπτικό μηχανισμό. Τώρα, το να μπούμε σε έναν τέτοιο μηχανισμό ως χώρα εκτός Ευρωζώνης σημαίνει ότι θα συμμετάσχουμε και στον ενιαίο μηχανισμό SSM. Και εδώ είναι τελείως διαφορετικοί οι κανόνες και αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Για ε, αυτή την πολύ δύσκολη πρόταση λοιπόν για την κατανομή των ψήφων σε home και host χώρες σας τονίζω ότι το συμφέρον των χωρών host μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό, τελείως διαφορετικό. Και επομένως να μην μπορεί να επιτευχθεί καμία συμφωνία. Αυτός ο κίνδυνος είναι σημαντικός. Νομίζω ότι οποιαδήποτε χώρα host στο Συμβούλιο Στήριξης θα πρέπει, ή επίλυση θα πρέπει να έχει κανόνες ανάλογους με εκείνους που ισχύουν στις χώρες home. Αν όμως δεχθούμε εδώ τους κανόνες που προβλέπονται για το SSM και προβλεφθούν κέρδη από διαμεθοριακές διευθετήσεις τότε πρέπει να ισχύει η αρχή ότι καμία χώρα δεν θα ζημιωθεί και καμία χώρα δεν θα φέρει μεγαλύτερο βάρος από τις άλλες. Έτσι δημιουργείται η αμφιβολία κατά πόσον έχει καλές προθέσεις εδώ η Κομισιόν. Εγώ δεν έχω ακόμη καταλάβει ποιες, πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις στο SRM. Οι δικαιοδοσίες που προβλέπονται θα ισχύουν μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά υπάρχουν, επαναλαμβάνω, χώρες εκτός Ευρωζώνης για τις οποίες προβλέπονται άλλες διαδικασίες ψηφοφορία. Θα θυμάστε τι είχε προβλεφθεί αρχικά. Αλλά οι τελικές συμφωνίες καταλήξαν πού. Οι προτάσεις της Κομισιόν εδώ στην ουσία διαγράφουν, απορρίπτουν τις προηγούμενες αποφάσεις. Μεχανισμού resolution. Rola EBC jako nadzorcy jest m.in. podejmowanie kroków zapobiegających powstaniu sytuacji. Εδώ υπάρχει και ο ρόλος της ΕΚΤ. Και θα καταλήξουμε ίσως στην αποτυχία οποιαδήποτε οποιοδήποτε μηχανισμού εποπτείας λόγω των θεσμικών διευθετήσεων που δεν μας επιτρέπουν ακόμη να καταλάβουμε αν ο στόχος είναι η στήριξη των τραπεζών ή η αποφυγή ανάληψης κινδύνου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Ζαντίκη. Yes, I apologize. I was voting in my other committee. ήμουν σε εργασίε άλλη επιτροπή. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και καθυστερημένα για την προστασία τη ενιαία αγορά και τι κρατικέ ενισχύσει. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι οι κρατικέ ενισχύσει, το σχετικό καθεστώ ισχύει σε όλο τον SRM. Ακόμη και αν ληφθεί μια υπόφαση από ένα υπερεθνικό οργανό και πάλι θα πρέπει να διέπεται από τους ε, κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε στους κανόνες όλη την ενιαία αγορά και επίσης για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό το δημόσιο χρέος ε, και Άκουσα την πρόταση να διαγραφεί αυτή η αναφορά στην κριτική ενίσχυση, κυρία Συγγήτρια, στην τροπολογία 28, ίσως έκανα λάθος, όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα ισχύουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και οι δύο λειτουργίες της Κομισιόν, δηλαδή ως ε, φορέα εξυγένσης, ε, σε αντίθεση με φορέα ανταγωνισμού θα πρέπει να διαχωριστούν. Διαφορετικά μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και νομίζω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον ε, ρόλο της Κομισιόν το μεταφύλακα του ανταγωνισμού. Επίσης, ε, χαίρομαι που διαγράφεται την δυνατότητα της Κομισιόν να μπορεί να πυροδοτήσει το μηχανισμό εξυγήνης από μόνη της, γιατί αυτό θα έθετε πολλά ερωτηματικά. Επίσης υπάρχουν ερωτήσεις σε σχέση ε, με το ρόλο της EBA, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών εκεί που έχουμε δώσει ρόλο διαμεσολάβηση στην NBA, τι σημαίνει αυτό για το ρόλο της Κομισιόν. Και χαίρομαι πολύ σκιώδες, συμφώνησαν ότι θα πρέπει ε, να μείνουμε κοντά στον νέο μηχανισμό εξυγίανσης. Ε, θα ήθελα να δω και σχέση σχέτιση του ενιαίου μηχανισμού εξυγένσης και τις οδηγίες για την ανάκαμψη και την εξυγένση, γιατί αν ε, αλλάξει κάτι στην ε, RRD, στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγένση, θέλουμε αυτό να αντικατοπτρίζεται και στον νέο μηχανισμό εξυγένσης, στον SRM. Πρέπει παράλληλα λοιπόν να οδεύουν τα δύο νομοθετήματα. Ξέρω ότι πολλοί αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι η πυροδότηση ε, του μηχανισμού δεν συνάδει, λέγονται στην έκθεση ΕΚΟΝ. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι αρμοδιότητες Μπέιλιν ε, ε, της Σερβία έχουν ε, ε ουσιαστικά εξελιχθεί και στην τροπολογία σας. σε σχέση με το θέμα της χώρας υποδοχής και της χώρας που φιλοξενείται ακούσαμε τους εκπροσώπους κάποιων χωρών που φιλοξενούνται και ανησυχώ για το άρθρο 51 και ο μηχανισμός ε, για την ψηφοφορία μήπως προσανολήθεστε πάρα πολύ στο κράτος υποδοχής και για το επίπεδο σχεδιασμού θα ήθελα και η ε, αρχές των χωρών φιλοξενούνται να έχουν κάποιες περαιτέρω αρμοδιότητες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Κομισιόν ε, να μπορεί να ανοίξει την πόρτα για κόστος ή για ευθύνες. Ε, δεν πρέπει να εκτίθεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κινδύνους στο μέλλον. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και τα εθνικά κοινοβούλια και θα πρέπει να υπάρχει και ευρωστή και νομίζω τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν και μόλις ακούσαμε τον Πολωνό συνάδελφο θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν. Και θα ήθελα μία διατύπωση που να ε, διασφαλίζει τι θα γίνει αν υπάρχουν κάποιες επιπλοκές. Πρέπει να έχουμε ασφάλεια δικαίου στο κείμενο. Και ξέρω ότι κάποιοι από τους συναδέλφους ανησυχούν γιατί σημαίνουμε πολύ αργό ρυθμό σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις για την Τραπεζική Ένωση. Όμως όλο αυτό δίνει ασφάλεια δικαίου στο όλο καθεστώς και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να βιαστούμε, να πάρουμε μια βιαστική απόφαση και τελικά να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου στο μέλλον, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν και από τον κατάλληλο δημοκρατικό έλεγχο. Φίλιππ, έχεις ζητήσει το λόγο ή όχι. Δεν θα σου ξαναδώσω το λόγο δεύτερη φορά Σβέν. Μπορεί να τα πει ο Φιλίπ αν θέλει. Συγγνώμη, προσπαθείς να δημιουργήσεις προηγούμενο εδώ. Όμως δεν πρόκειται να υποχωρήσω. Αν δεν υπάρχει κανένας καινούριο να πάρει το λόγο, θα ξαναδώσω το λόγο στην συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά για να είμαι πιο γρήγορη. Γιατί έχουμε καθυστερήσει κάπως. Δεν θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους όσους μίλησαν. Αλλά να σας ενημερώσω ότι σημείωσα δεόντως όλα τα σχόλια και τις προτάσεις και θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ στο δυνατό περισσότερο αυτό το καλό πνεύμα συνεργασίας που νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί. Είμαι πολύ ευαίσθητη απέναντι στην ανάγκη να δημιουργήσουμε το BRD ως ένα πλαίσιο και να το καταστήσουμε πλήρως ε, συμβατό με τον SRM, τον νέο μηχανισμό Τον έχουμε τον SSM και τον SRM. Η δική μου ερμηνεία και νομίζω πρέπει να μείνουμε εκεί είναι πολύ κοντά στην περιγραφή της Μαριαν Τίσεν. Δηλαδή, φυσικά καλύπτονται οι τράπεζες από αυτό, αλλά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και στα κρατή-μέλη, για ποιες ε, τράπεζες υπάρχει ενιαία εποπτεία και μια εξυγίανση, γιατί διαφορετικά δεν θα έχει νόημα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως αν έχουμε μια ισχυρή εποπτική αρχή, τότε άμεσα ή έμεσα έχει πλήρες εξουσίες για τις τράπεζες που εδρεύουν σε κάποια κρατημέλη και κατόπιν είναι αναπόφευκτο να έχουμε ένα κοινό μηχανισμό εξυγίασης Όλα αυτά θα πρέπει να οδεύουν από κοινού και να μην έχουμε και ροχμές στην εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι είναι κρίσιμη ισορροπία και θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Η δεύτερη πτυχή αφορά τα διάφορα σκέλη της δομής. Εδώ. Λυπάμαι που ο συνάδελφος Πίτερ Σάιμον δεν είναι πια εδώ γιατί νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι έχουμε το σύστημα εγγύσεις καταθέσεων και την κοινή εποπτεία και το ότι θα έχουμε ένα κοινό, ένα νέο μηχανισμό εξυγίανσης, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι τρεις πυλώνες έχουν διαφορετική σημασία για την Τραπεζική Ένωση, γιατί έχουμε ενιαία εποπτική ορχή, θα έχουμε και μια ενιαία αρχή εξυγίανσης και έναν ενιαίο μηχανισμό και ένα ενιαίο τομείο, αλλά σε ό,τι αφορά την εγγύηση των καταθέσεων έχουμε συστήματα μεμονωμένα. Επομένως, δεν υπάρχει συνεργασία που να έχει καθοριστεί εκ των προτέρων σε ό,τι αφορά την ασφάλιση των καταθέσεων των πολιτών που είναι υπό την κοινή εποπτεία και την κοινή εξυγίανση. Έτσι λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το έχουμε ξεκάθαρα στο νου μας και θα προστατεύσουμε μόνο τις καταθέσεις επιστρέφοντάς τις αν προκύψει η τελευταία περίπτωση μέχρι τις 100.000. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα έχουμε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που θα προσφέρει σαφήνεια για το πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με το μέσο του Μπέιλιν. Φυσικά, έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να έχουμε ένα κοινό Μπέιλιν, να έχουμε δηλαδή κάποιους κοινού κανόνες και κατόπιν πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση για το πότε τα διάφορα ταμεία εξυγίανσης ή το νέο ταμείο αναλαμβάνουν δράση και επίση αυτό είναι και ο ρόλος αυτού του Ταμείου Εξυγένσης και εγώ δεν ε, βλέπω ότι το Ταμείο ε, είναι ένα Ταμείο που πληρώνει, επιστρέφει τα χρήματα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας μηχανισμός κεφαλαϊκός που θα μας βοηθήσει να εξηγιάνουμε ένα ίδρυμα. Και επίση όλε οι καταθέσει δεν είναι το ίδιο. Καταλαβαίνω ότι μεγάλε καταθέσει δεν μπορούν να τυχούν τη ε, ίδια μεταχείριση όπω οι καταθέσει των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν ελπίζω να βρούμε μια κοινή προσέγγιση γι' αυτό, αλλά δεν θα μπορέσω να εξηγήσω στους πολίτες ότι έχουμε ένα ταμείο που θα μπορεί να διασφαλίζει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία για τις καταθέσεις θα έχουμε μόνο το Εθνικό Μηχανισμό Οικονομικής Στήριξης για να αποπληρώσει τις καταθέσεις μέχρι τις 100.000. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Φυσικά, αναγνωρίζουμε την ύπαρξη των ε, συστημάτων προστασίας, των Εθνικών Συστημάτων Προστασίας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα συστήματα, αλλά θα πρέπει να αγγιθούμε και στους άλλους πολίτες, σε άλλες χώρες που δεν εντάσσονται στα συστήματα αυτά. Όχι 100% ίδια προστασία, αλλά να τους δώσουμε κάποιες εγγύσεις. Και κατόπιν έχουμε το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε πως αυτό το ταμείο θα πρέπει να ενισχυθεί για να ξεκινήσει με κάποια αξιοπιστία. Φυσικά όλοι εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο για να εγγυηθούμε ότι το Ταμείο δεν είναι ένας χάρτινος τίγρης. και θα χρειαστεί αρκετός καιρός ε, για να καταστεί εύρωστο χρηματοοικονομικά. Έτσι λοιπόν, πραγματικά θα ήθελα να λάβω κάποιες συνεισφορές σχετικά. Κατανοώ ότι αυτό το πρόβλημα άρχισε να είναι ζήτημα και στο Συμβούλιο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή διατύπωση που θα επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Σημείωσα και το πρόβλημα με τις ε, εξουσίες ψήφου. μέσω της ε, παρουσίας των κοινωτικών θεσμών, των κοινωτικών οργάνων θα πρέπει να εγγυηθούμε κάποιο κοινό πολιτισμό, κάποια κοινή προσέγγιση σε σχέση με το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις των διάφορων εκτελεστικών συμβουλίων. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε αυτό. Σημείωσα και το αίτημα της κυρίας Βορτμαν Κόλ, αφενός, αφετέρου. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς ποιο ήταν το μήνυμα της Σιλβή, αλλά κατάλαβα ότι ήταν κάπως πιο διστακτική να δώσει δικαίωμα ψήφου στην ΕΚΤ. Θα πρέπει να το λύσουμε λοιπόν και αυτό. έχουμε πολλά ζητήματα βέβαια, αλλά από ό,τι κατάλαβα συμφωνούμε σε σχέση με το ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο το ποιο πυροδοτεί το πότε ένα Ίδρυμα μπαίνει σε στάδιο εξυγίανσης, αλλά θα πρέπει να επιλύσουμε και άλλα θέματα που προς το παρόν δεν έχουμε συζητήσει. Ένα από αυτά ε, ήταν ε, το θέμα της μετάβασης, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κλίν. Και μιλάμε για την μετάβαση όχι για το τι θα γίνει με τα εθνικά ταμεία εξηγήνσης που ήδη υπάρχουν, αλλά ε, τι θα γίνει και με τη λειτουργία του συστήματος. Και ένα εγχειρίδιο, ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων σε ό,τι αφορά την ανακεφαλοποίηση τη λειτουργία των ταμείων. Πολύ σαφείς και συνάδελφοι, όπως και η κυρία Μπόλς, σε αυτό κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την προληπτική κεφαλοποίηση που προτίθηκε στην BRRD από το Συμβούλιο που μπορεί να γίνει επικεφαλοποίηση από εθνικά κονδύλια εκ των προτέρων. μέσω παραδείγματος χάρη της ε, Συμφωνίας επί των Αρχών των Εισηγητών. Πώς ε, θα γίνει αυτό στα πλαίσια του ενιαίου μηχανισμού εξυγένσης και του ενιαίου μηχανισμού υποπτίας. Υπήρχαν και άλλα θέματα. Προσπάθησα να σημειώσω όλες τις συστάσεις που ακούστηκαν και από την κυρία Λούλινγκ θα πρέπει να λειτουργούμε πάρα πολύ ξεκάθαρα για το πώς ε, αντιμετωπίσουμε το θέμα των σχέσεων μεταξύ των μελών των τραπεζών που βρίσκονται εντός της Τραπεζικής Ένωσης και αυτών που θα είναι εκτός. Αλλά ένα τμήμα αυτού προέρχεται κατευθείαν από την BRRD και όχι από τον SRM. Νομίζω ότι είναι γεμάτο προκλήσεις το κείμενο. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες επί των άρθρων. Που έχουμε και συγκεκριμένε ερωτήσει που τέθηκαν από το Σβέν και από τη Βίκη Φόρτ. Νομίζω ότι υπήρξε μια αλλαγή και στα νούμερα. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος των τροπολογιών των δικών μου ήταν ε, να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες, όπως ε, το ερμήνευσε ακριβώς και η κυρία Φόρτ, να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες σαν η αρχή εξυγίανσης λάβει μια απόφαση που δεν ε, ερμηνεύεται όπως πρέπει από την Εθνική Αρχή Εξυγίανσης, τότε υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Όταν λοιπόν βάζουμε, αν βάλουμε αυτές τις τροπολογίες στο σωστό πλαίσιο, γίνεται πιο σαφές. Και σε σχέση με την εθνική συμμετοχή, ο δικός μου στόχος μεταξύ, μέσω των διάφορων τροπολογιών είναι ότι δεν μπορούν οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο κοινωνικό επίπεδο που να έχουν ε, άμεση ε, συνέπεια στην ε, φορολογικές δημοσιονομικές οξύες των κρατών μελών αλλά αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι εννοώ στους συναδέλφους σε προσωπική βάση και να αναδιατυπώσω. Σας ευχαριστώ, έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Θα δω πολύ προσεκτικά όλες τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων και σας ευχαριστώ για αυτή την ανοιχτή συζήτηση. Με βοήθησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ πολύ. 18 Οκτωβρίου λίγη διορία κατάθεση τροπολογιών, είχε αναγγελθεί εν καιρός. και είχαμε ανοίξει τη διορία αμέσως μόλις κατατέθηκε η έκθεση. Το μάθαν όλοι εγκαίρως. ...18 Οκτωβρίου λοιπόν λίγη στις 5 το, μεσή, το απόγευμα και στις 18 Νοεμβρίου η συζήτηση ψηφοφορία στην εικόνη 25 Νοεμβρίου και Ολομέλεια τον Μάρτιο του 14 ελπίζοντας βέβαια να έχουμε έρθει σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Και τώρα το επόμενο θέμα που είναι που είναι Α, ναι, ναι, ναι, ναι, Είναι συζήτηση των τροπολογιών για την έκθεση του Hans Peter Martin, ο οποίος όμως λείπει γιατί είναι στο ίδιο συγκοινωνιακό πρόβλημα στο οποίο βρίσκονται και άλλοι πολλοί σήμερα και γι' αυτό θα διαβάσω εγώ εξ του εισηγητού για την γνώμη χορήγηση και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από και δραστηριότητε που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτό τη Ένωση. Τελεία. Λοιπόν, καταρχήν ζητώ συγγνώμη, λέει ο Χάνς Πίτερ, γιατί υπήρξε ένα δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία και έκλεισε τελείως. Ευχαριστώ όλους τους κοιότης που έχουν συνεργαστεί μαζί μου τόσο θετικά, μαζί με του τους όλων των πολιτικών ομάδων και καταλήξαμε σε λογικούς συμβιβασμούς. Έχουν ζητηθεί δύο ψηφοφορίε σε τμήματα για τους συμβιβασμούς Γ και Ήτα, αλλά ε, η θέση μου είναι να τους δεχτούμε. Γενικά είμαι ικανοποιημένος γιατί μπορέσαμε να δεχτούμε σημαντικά να συμφωνήσουμε για σημαντικά σημεία όπως για τους παραλήπτες των σχεδίων της ΕΤΕ κλπ. Και επετεύχθη επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια της χρηματοδότησης από την ΕΤΕ. Ταυτόχρονα μειώσαμε, καταφέραμε να μειώσουμε την κερδοσοκοπία. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα οι σκιώδεις και οι άλλοι να σχολιάσουν τις τροπολογίες και ο Χάνς Πίτερ Μάρτιν ελπίζει να έρθει σήμερα, αν και δεν κατάφερε μέχρι τώρα. Τέλο πάντων, αυτά μου είπε να δηλώσω. Δεν ξέρω αν κανένας από τους σκιώδεις θέλει να σχαλιάσει. Ο κύριος Λούχαν μήπως. Ναι, ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Στόλογιανό Σκιώδη. θέλει μερικές αλλαγές μετά από συζήτηση με βουλευτές του ΕΛΚ. Θέλει ψηφοφορία σε τμήματα για τη συμβιβαστική γάμα. Ε. Ε, with, um, with a που μιλάει για την προοδευτική απόσβεση μέχρι το τέλος σε δύο τμήματα λοιπόν χωριστή ψηφοφορία στο ΕΛΚ τα συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και δεν βρίσκουμε λογικό οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες να προτιμούνται γιατί υπάρχουν μερικές χώρες που εξαρτώνται από τους παραδοσιακούς ενεργειακούς πόρους και δεν πρέπει να τις εμποδίσουμε να αναπτυχθούν. Αυτό είναι το επιχείρημα. Άλλη τροπολογία για τη συμβιβαστική ή τα σημεία 14 του σκεπτικού και εδώ ζητάμε ψηφοφορία χωριστή και σε τμήματα. Χωριστά την τελευταία φράση δηλαδή που μιλά για αποκεντρωμένα προγράμματα ανανεωσίμων. Δεν είναι βέβαια τώρα η καταλληλότερη ώρα να θέσουμε τις προτεραιότητες, αλλά υπάρχουν μερικές χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα και δεν πρέπει να απαιτούμε αυτά που απαιτούμε από τις χώρες αυτές. Λοιπόν, χωρίς ψηφοφορία για τη συμβιβαστική ήττα, μετά αποσύρουμε την τροπολογία 78 που είχε γραφτεί από τον κύριο για τον ίδιο. Is already on the Να, αυτά είναι που ήθελα να σας πω βασικά. βασικά. Και ευχαριστεί και όλους τους σκιώδεις και μη σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία και χαίρεται που φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο. Γιατί μέχρι τώρα ήταν πολύ αφιλεγόμενο το θέμα μέχρι και την περασμένη εβδομάδα στο ΕΛΚΑ αλλά τώρα εντάξει και αυτά δεν, είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ευχαριστώ. Όχι, ε, όχι. Έχουμε και άλλες δύο προφορικές τροπολογίες των φιλελευθέρων. Α, είναι από πίσω η φιλελεύθεροι. Εντάξει, καλά, ναι, εντάξει, ναι, καλά. Τώρα, εκ μέρου των ε, σοσιαλιστών, Ελίζα, εσείς ε, θα εκπροσωπήσετε τον κύριο Μπέρμαν. Ναι. Εκ μέρους του λοιπόν ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέταξαν την έκταση και πράγματι η ομάδα των σοσιαλιστών στηρίζει ανεπιφύλακτα τις ε, προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Η πρόταση της Επιτροπής είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι η νέα απόφαση οδηγεί τις δραστηριότητες της ΕΚΤ σε κοινωνικούς τομείς που συνδυάζουν καλύτερα την πολιτική της ΕΚΤ με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, για μας είναι πολύ σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο θέμα της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην κλιματική αλλαγή, τόσο όσον αφορά την άμπλυνση των φαινομένων, όσο και την προσαρμογή. Επίσης, είναι σημαντικό το ότι στην πρόταση αναφέρεται η εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την επόμενη περίοδο από το 14 το 20 με πιθανότητα εξαμήνου παράτασης έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΚΤ και αυτό είναι καθοριστική σημασία. Πρόκειται λοιπόν και πάλι για το εξή. Ε, ε, το σχέδιο της γνωμοδότησης βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα εμάς μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε τη ζήτηση και να μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, τις πρακτικές να τις συνδυάζει με το μακροπρόθεσμο μέλλον χωρίς να γίνεται ε, ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των φορολογικών παρδίσεων. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, να είναι πιο διαφανής όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προσφέρει, για να ξέρουμε πού κατευθύνονται τα κονδύλια. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα της ε, διαφάνειας και του σεβασμού όλα αυτά που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε με τους ε, ε, φορολογικούς ε, παραδείσους και συγκεκριμένες νομοθεσίες, εμείς στηρίζουμε τις συμβαστικές προτάσεις και για άλλη μια φορά ευχαριστούμε τον συντάκτη για την γνωμοδότησή του. Αυτή, αυτό μονέθεσε να σας πω. Ο Νίλς εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Σε γενικές γραμμές ε, στηρίζουμε τις συμβαστικές που προέκυψαν από τη συνάντηση των σκιωδών. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά για τη διαφάνεια και το ε, πλήσιμο, ε, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έτσι λοιπόν εγώ Προτείνω δύο τροπολογίες. Η μία είναι να διαγραφεί ένα τμήμα του 74 και η άλλη ε, τροπολογία 16. Αυτά τα έκανα σε συνεργασία και σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προτείνω σε αυτό το άρθρο να διαγράψουμε το αίτημα που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, θα πρέπει να διακόψει τη ροή χρηματοδοτήσεων μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να ε, ανασταλεί η εκταμίευση ε, όσο τρέχει η, τρέχουν ανακρίσεις. Αυτό ε, πράγματι απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι πολιτικές για τις απάτες και τη διαφθορά αυτό ισχύει και για τις ίδιες τις έρευνες της Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης η Τράπεζα λέει ότι οι διατάξεις είναι σε επίπεδα αγοράς και είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει ε, να είναι ούτε προς το συμφέρον της Τράπεζας Επενδύσεων ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το να ξαναρχίσει η έκθεση από την αρχή. Γι' αυτό προτείνουμε ε, προφορική τροπολογία σε αυτό το άρθρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως θέλει κανείς να εκπροσωπήσει τους πράσινους επί του θέματος. Ε, κοίταξε, είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το να μιλάω εξ ονόματος κάποιου που δεν είναι εδώ και να απευθύνουμε σε κάποιον που ούτε και αυτός είναι εδώ. Τέλος το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα στηρίξουμε όλες τις ε, σημαστικές προτάσεις του εισηγητή. Να πω μόνο το εξής. Άκουσα τι είπε ε, κάποιος που και αυτός δεν είναι εδώ, ο Στόλογια, δηλαδή ότι δεν θα πρέπει να περιορίσουμε τη χρηματοδότηση μόνο σε προγράμματα ε, που να βρίσκονται στον ενεργειακό τομέα και στις ανανεώσιμες πηγές. Θέλω να πω ότι αυτό ε, που χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι τεχνολογία του προηγούμενου αιώνα και όχι του επόμενου ή αυτού του αιώνα. Και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι τα νέα κρατεμέλη δεν ενδιαφέρονται και δεν είναι επιλέξιμα το δυναμικό ε, ηλιακής ενέργειας και ολικής ενέργειας σε αυτές τις χώρες είναι το ίδιο όπως και στις υπόλοιπες χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό αυτό που λέτε εγώ δεν το δέχομαι. Κάτι άλλο το οποίο θα προχωρήσουμε, αν και είμαστε μειονότητα, ε, για μια φορά συμφωνούμε με την κυρία Λούλινγκ. Όπως σας είπα, το γεγονός ότι η BRD θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί πια δεν θέλουμε να υπάρχουν άχρηστοι θεσμοί. Όλα αυτά ε, κοστίζουν χρήματα και ε, δεν συνεπάγονται τίποτα το θετικό. Κανείς άλλος παρακαλώ. Υπήρξαν 78 ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν συμπεριλαμβάνουν αυτών και του εισηγητή. Η άποψη της ε, οίκων ε, πλέον έχει διαμορφωθεί και θα ψηφίσουμε σήμερα διότι η κύρια επιτροπή, η Επιτροπή Προπολογισμού θα ψηφίσει σύντομα και θέλουμε να συμπεριλάβει και τη δική μας την άποψη. Γι' αυτό λοιπόν προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχει κανείς σας τα... τις τροπολογίες. Τις έχετε μπροστά σας. Για να δούμε αν μπορούμε να ψηφίσουμε ε, χωρίς ε, κάρτες. So Right. So uh, all... Ωραία. Υπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. 13. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Δεν ε, είστε και πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας γιατί διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα. Τροπολογία 14, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 47, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός α, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γάμα σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές, κάπως παραξενώ το αποτέλεσμα μπορείτε να μετρήσετε πιστεύετε Θα μετρήσει η γραμματεία. Πώς είστε υπέρ, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι. Υπέρ. Περιμένετε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα του συμβασμού C. Και πρέπει να μετρήσουμε, θα ψηφίσουμε ένα σχηρός. Παρακαλώ υπέρ. Μάλιστα, το κάνουμε ηλεκτρονικά, λέει η Πρόεδρος. Wait whilst I find a card now. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Δεύτερο τμήμα του Ψήφισατε όλοι. Μάλιστα, γκρίνεται 16 υπέρ, 11 κατά. Περνάμε στην 52 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. 52. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 10 με 17. 53 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά εποχές θα ελέγξουμε την 54. τε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται, να το ελέγξουμε όμως. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η είναι την προηγούμενη. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε νομίζω ότι εγκρίνεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται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 Μπερδεύτηκα. Για την 66 υπέρ. Κατά. 66 σαν πόλ. Είσαι υπέρ ή κατά. Είσαι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός D. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 με προφορική τροπολογία της Άλντε. Είναι όλοι ικανοποιημένοι με την προφορική τροπολογία, δεν υπάρχει αντίρρηση. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 78 έχει αποσυρθεί πάμε στο συμβασμό F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνδεσμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνδεσμός H σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 καταπίπτει, 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 33 παρακαλώ. το όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 37. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ 16 κατά 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σαρανταένα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 42 υπέρ, κατά σε εγκρίνεται 43 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά σε εγκρίνεται 44 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε τη 44 γιατί ήρθαν και άλλοι Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στο συμβασμό I υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 11. Συμφωνείτε με την προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για όλο το κείμενο που τροποποιήθηκε έρχεται η ψηφοφορία. Θα κλείσω την ψηφοφορία. Πέρας. 32 υπέρ. Κανείς κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Η επόμενη συνεδρίασή μα. θα είναι στι 17 Οκτωβρίου στι 9 το πρωί. Σα ευχαριστώ.